Να ξαναρχίσουμε λοιπόν τις εργασίες της Επιτροπής μας ε, λέγοντάς σας ως ε, ήθιστε ότι μεταδίδονται, ε, μεταδίδονται από την εσωτερική τηλεόραση και από το διαδίκτυο οι εργασίες μας. Η Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, η κυρία Γουόλη, την οποία θερμότατα καλωσορίζουμε, θα μας μιλήσει για τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το κοινό Μητρό Διαφάνειας. Η κυρία Γουόλης ήταν πρόεδρος της ομάδας εργασίας που διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία και η οποία ενεκρίθη από την 18η Δεκεμβρίου από τη διάσκεψη των Προέδρων. Νομίζω ότι κατά την άποψή μου μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις. Θα πρέπει να πάρουμε δύο αποφάσεις. Μία η οποία αφορά την έγκριση της συμφωνίας την, ε, οι για την τροποποίηση ε, της ε, συνθήκης γιατί θα πρέπει να τροποποιηθούν τα σχετικά άρθρα. Η κυρία Γουόλης όμως από το ύψος των γνώσεών της θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γουόλης που ήρθατε για το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και που με καλέσατε στην Επιτροπή σας σήμερα και για την ε, συνεργασία σας στη δουλειά αυτή. Έχετε μπροστά σας, συνάδελφοι, το σχέδιο της διαθεσμικής συμφωνίας μεταξύ ημών του Κοινοβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό μητρό διαφάνειας, όπως αποκαλείται. Έχετε λοιπόν μπροστά σας τα έγγραφα. Να πω ίσως δύο λόγια καταρχάς για το ιστορικό υπόβαθρο της υπόθεσης αυτής. Βρισκόμαστε στο σημείο αυτό σήμερα με την Επιτροπή σας για να ξεκινήσουμε τις ε, κοινέ διαβουλεύσεις για το κοινό Μητρό Διαφάνειας λόγω μια έκθεση την οποία συνέταξε η Επιτροπή σας την προηγούμενη θητεία. Αλεξάνδρου Στουτ ήταν ο εισηγητής και ο κύριος Φρέντριχ τη συνέχισε για την θέση των εκπροσώπων συμφερόντων, των εκπροσώπων λόμπι και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν γέννη από τα θεσμικά όργανα. Η έκθεση αυτή παρουσίασε την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα εργαστίας η οποία θα δημιουργηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων, κυρίως μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιστροπής, για να δημιουργηθεί ένα κοινό μητρό. Και αυτό ήταν λοιπόν το έργο το οποίο ξεκινήσαμε, ξεκίνησε την προηγούμενη θητεία, η εργασία αυτή, υπό τη δική μου ηγεσία και συνεχίζει και ολοκληρώνεται στην τρέχουσα θητεία. Ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κασίνη, ο κύριος Γεωλάιναν, ο οποίος ήταν ο προ... προηγούμενος πρόεδρος της Επιτροπής, συμμετείχαν στις εργασίες αυτές και η κυρία Ντουρά. Εκπροσωπούνταν λοιπόν όλες οι βασικές ομάδες ε, του Κοινοβουλίου. Αρχικά μιλούσαμε με τον Σιμ Κάρλος ε, και τον Μάριο Σεύκοβιτ, την τρέχουσα θητεία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τη συμφωνία, την οποία ε, πετύχαμε. Καταρχά, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διατύπωση, για να ξέρουμε τι συζητάμε δεν μιλάμε πλέον για τους εκπροσώπους συμφερόντων, μιλάμε στον τίτλο για Μητρό Διαφάνειας. Θα σας εξηγήσω γιατί καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε τους συγκεκριμένους όρους. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αντιλαμβανόμαστε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της προηγούμενης θητείας, το οποίο ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο θα ήθελε να υπάρχει ένα υποχρεωτικό μητρό για όλους εκείνους που προσπαθούν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι υποχρεωτικό μητρό, θα το ξέρετε αυτό, γιατί όπως ξέρετε πιο πολλοί από εσάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα εθελοντικό, εθελούσιο μητρό. Είναι λοιπόν αντίθετο αυτό με αυτό που θέλει το Κοινοβούλιο. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, να εκφράσουμε ότι ο απότερος στόχος του Κοινοβουλίου είναι ένα υποχρεωτικό μητρό. Καταλαβαίνουμε βέβαια και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που μπορούμε να πετύχουμε στην παρούσα φάση είναι ίσως ε, ένα ασφαλές εθελούσιο μητρό. Και αυτό ε, κάτι σημαίνει γιατί για παράδειγμα οι εκπρόσωποι των ε, συμφερόντων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν μια κάρτα για να μπουν στο κοινοβούλιο. Πολλά έχουμε αναφέρει υπέρ του υποχρεωτικού χαρακτήρα του Μητρώου και πολλοί εκπρόσωποι συμφερόντων μας αναφέρουν ότι και αυτοί δεν το προτιμούσαν να είναι υποχρεωτικό, αλλά η νομική γνωμοδότηση ήταν σαφής προκειμένου να είναι υποχρεωτικό το μετρό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο του, της συνθήκης το οποίο απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Στην παρούσα φάση λοιπόν, αν και το κοιτάμε, περιοριζόμαστε και συζητάμε τη δημιουργία ενός εθελοντικού μητρώου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, αυτό που πάντα ήταν σαφές στο μυαλό μας είναι ότι ασφαλώς υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον τρόπο, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του ο Ευρωβουλευτής, ο κάθε Ευρωβουλευτής. Δεν θα πρέπει αυτό να αποτελέσει εμπόδιο στην ελεύθερη ε, διακίνηση, στην ελεύθερη ε, λειτουργία των Ευρωβουλευτών. Αυτό είχαμε λοιπόν υπόψη. Και προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα του αυτού. Σκοπός είναι οι πολίτες μας να εμπιστευτούν, ελπίζουμε, πιο πολύ την ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων, να καταστήσουμε σαφές ότι να καταστήσουμε σαφές ποιος μας μιλάει για την ευρωπαϊκή πολιτική, ποιος επηρεάζει την ευρωπαϊκή πολιτική μέσω του Μητρώου Διαφάνειας. Να οικοδομήσουμε λοιπόν μια εμπιστοσύνη με τους πολίτες σε ό,τι αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων και φυσικά να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διάφορων φορέων που εμπλέκονται. Ένα από τα θέματα το οποίο παρουσίασε δυσκολίες εκ πρώτης όψεως και γι' αυτό λοιπόν δικαίως καταλήξαμε στο Μητρό Διαφάνειας όπως αποκαλείται είναι το εξής πολλά άτομα που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι, δεν ε, αρέσκονται στον όρο λόμπι. Δεν τους αρέσει να χρησιμοποιείται ο όρος λόμπι για αυτούς. Θέλουμε λοιπόν να είναι όσο πιο, δυνατόν, πιο ευρεία δυνατόν η κάλυψη του Μητρώου αυτό. Και θέλουμε ο κόσμος να χαίρεται που συμμετέχει και που εγγράφεται στο Μητρώο αυτό οι βασικοί εμπορικοί φορείς, αυτοί που πραγματικά εκπροσωπούν συμφέροντα είναι λομπιίστες εμπορικοί, είναι η πρώτη και μιλήσαμε πάρα πολύ με τους ε, νομικούς για να διευκρινίσουμε τις διαφορές αυτές και θα πρέπει να διακρίνουμε τους εκπροσώπους συμφερόντων με, τον, με τους εκπροσώπους τους εμπορικούς. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι όλες οι κατηγορίες θα συμμετάσχουν στο Μητρό και θεωρώ ότι θα είναι τεράστια επιτυχία σε ό,τι αφορά την συμμετοχή πολλών ομάδων, πολλών οντοτήτων στο Μητρό. Βλέπετε ότι από το τρόπο που διαμορφώνεται το Μητρό Έχουμε τις εμπορικές ε, οντότητες και έχουμε και τις λοιπές οργανώσεις. Αυτό καθησύχασε τους πάντες και προσπαθούμε λοιπόν να επιλέξουμε τη λέξη διαφάνειας, να μην μιλάμε για λόμπι το οποίο αναστατώνει αρκετούς. Να πούμε δύο λόγια για το περιεχόμενο του Μητρώου. Ήταν σαφές ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πιο πολλές ε, πληροφορίες που για τα άτομα που καταχωρίζονται σε ό,τι αφορά το, το χρηματοπιστωτικό τους καθεστώς. Μετά από τα χρόνια που τηρεί το Μητρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι έχει εμπειρία και θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος. Αυτό νομίζω λειτουργεί πολύ καλύτερα θα υπάγεται σε ένα κοινό κώδικα διοντολογία στο Μητρό για τις σωστές διαδικασίες. Αν λάβουμε κάποια ε, καταγγελία ε, θα μπορέσει να ελεγχθεί και από τα δύο θεσμικά όργανα και αν φυσικά αντιληφθούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην διαδικασία φυσικά μπορεί να γίνει και καταγγελία στον διαμεσολαβητή. Υπάρχει λοιπόν ένα πλήρες σύστημα το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και να ικανοποιήσει τους πάντες, όπως ελπίζω. Για το Κοινοβούλιο, το ότι πετύχαμε ένα κοινόμητρο με την ε, Επιτροπή, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ένα θέμα εσωτερικής διαχείρισης. Το σύστημα με το BATS, για παράδειγμα, Γι' αυτό δώσαμε ένα, ένα μεγάλο περιθώριο στον εαυτό μας για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία το όλο σύστημα. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα πολύ σωστά και θα πρέπει να γίνουν οι διαδικαστικές αλλαγές μέσω της Επιτροπής εδώ. Το ίδιο θα γίνει και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους εσωτερικούς τους κανονισμούς. Αυτό λοιπόν το ιστορικό υπόβαθρο, αυτά περάσαμε ως ομάδα εργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι τελικά το αποτέλεσμα είναι σωστό. Ελπίζω και εσείς να συμφωνείτε μαζί μου. Και ελπίζω να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τη διαθεσμική συμφωνία και ενδεχόμενε αλλαγές για το ιστορικό μας κανονισμό. Θα θέλαμε το κοινό μητρόνο να λειτουργεί μέχρι τον Ιούνιο και να επάγεται. Φυσικά ε, υπό τον όρο ότι θα εγκριθεί από την Επιτροπή σας, θα ήταν καλό να τηρηθεί αυτή η προθεσμία και θα πρέπει να πω ότι το κοινό μητρό θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Συμβούλιο. Λάβαμε μία σειρά πρωτοβουλειών στην τρέχουσα θητεία για να συμπεριλάβουμε και το Συμβούλιο. Και ήταν θετική η αντίδραση από τη Βελγική Προεδρία έγινε και μια σχετική συνάντηση την περασμένη εβδομάδα. Ήταν ακόμα πιο θετικό το μήνυμα που λάβαμε. Συνεχίζονται οι συζητήσεις λοιπόν και μπορεί μέχρι τον Ιούνιο να βρεθούμε στην κατάσταση όπου θα έχουμε ένα μητρό το οποίο θα περιλαμβάνει και τα τρία θεσμικά όργανα, το οποίο ασφαλώς είναι και ευκταίο. Αυτά λοιπόν επιγραμματικά τα γεγονότα και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, αλλά εσείς ασφαλώς είσαστε οι δήμονες στα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γουόλης για την ε, εισήγησή σας και θα δώσω τώρα αμέσως τους συναδέλφους, πρώτος εκ των οποίων έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Ντάφ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την συνάδελφό μας για την εξαιρετικά επαγγελματική προσέγγιση που έκανε στο θέμα, καθώς επίσης και για την εξαιρετική παρουσίαση της ε, πρόοδου ε, που έχει λάβει χώρα στο θέμα. Υπάρχει πρόοδος. Υπάρχουν όμως ακόμα και κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να διαλευκανθούν Ήταν ε, προτίμησή μας να έχουμε υποχρεωτικό μητρό και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να επιβάλλουμε την άποψή μας. Εάν ε, βάσει του παλαιού μηχανισμού Ε, βάσει του άρθρου 395 αν δεν κάνω λάθος. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει δηλαδή μέσω του 395 ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει μέσω κανονισμού. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένω την απόφαση της νομικής υπηρεσίας και την αιτιολόγησή της γιατί απαιτείται ε, εν προκειμένου στο Συμβούλιο ε, ομοφωνία για ένα τέτοιο θέμα. Έχουμε εμπειρία από παλαιές γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας που κατά την άποψη της Επιτροπής μας ε, είχαν μάλλον εσφαλμένη πορεία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ε, δω πρόοδο, σαν αυτή που ανέφερε η Διάννα Γουόλους ότι υπάρχει σε σχέση με το Συμβούλιο. Um, Έχω την εντύπωση, μάλλον μου δημιουργήθηκε η εντύπωση, ότι οι εγγεγραμμένοι είναι ικανοποιημένοι από την ε, διαδικασία, αλλά ε, θα θέλαμε να ε, πάμε ακόμα παραπέρα. Βλέπω πολύ συχνά στο έγγραφο την έκφραση expected to be registered που αναμένουμε ότι θα καταγραφούν. Διαβάζω εδώ μια συγκεκριμένη παράγραφο, ας πούμε, προτείνεται οι οργανώσεις των εκκλησιών ε, αναμένεται οι οργανώσεις των εκκλησιών να καταγραφούν. Αλλά ε, δεν ε, αφορά τις εκκλησίες τις ίδιες αυτό το Μητρό. Αναρωτιέμαι αν μπορεί η κυρία Γουόλης να μας το εξηγήσει λίγο καλύτερα αυτό. Πάντως, στο σύνολο θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε πρόοδο. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε κάποιες αναθεωρήσεις τους δικούς μας κανόνες λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Γκρότε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Αντιπρόεδρό μας. Νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στο θέμα της διαφάνειας. Γιατί κάθε ομάδα επισκεπτών, κάθε ομάδα επισκεπτών ε, Ξέρετε, αναφέρεται ότι α, είναι ελεύθερο, α, ελεύθερη η πρόσβαση εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιος θέλει μπαίνει, ποιος θέλει βγαίνει. Ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ καλό αν καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το κοινό μητρό διαφάνειας και χαίρομαι που το αναφέρατε ότι για να είναι εκείνο το Μητρό χρειάζεται και το τρίτο θεσμικό όργανο. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό όργανο και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ακούμε ότι και το τρίτο όργανο ε, αναλογίζεται να συμμετάσχει στο κοινό Μητρό. Το σημαντικό στοιχείο είναι να υπάρχουν πειθαρχικέ ε, δυνατότητες, δηλαδή αν υπάρχει κάποια τεράστια παραβίαση. Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε, να υπολογίζουμε σε συνέπειες για αυτούς που έκαναν την παραβίαση του Μητρώου και, όπως είπε και ο συνάδελφος Ντάφ πριν από λίγο, δεν θα πρέπει να είναι εντελώς εθελοντικό το Μητρό. Θα πρέπει να επισέλθουν όσο πιο πολλά υποχρεωτικά ε, στοιχεία γίνεται. Γιατί ένα πράγμα με έχει εντυπωσιάσει στην πολιτική. Ξέρετε, ό,τι ε, δεσμεύσει αναλαμβάνονται σε θελοντικό επίπεδο, ε, σε μεγάλο επίπεδο αμελούνται. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό να υπάρχει διαφάνεια υποχρεωτική. Έχουμε μια μεγάλη σειρά ομάδων ε, εκπροσώπων συμφερόντων που έχουν πρόσβαση εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 20 έως 30.000 αναφέρεται το αριθμητικό στοιχείο το σχετικό. Είναι τεράστιος ο αριθμός αυτός και θεωρώ λοιπόν ότι για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι ένα καλό μήνυμα να υπάρχει δεσμευτικό σύστημα και να είναι το σύστημα αυτό ένα σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει και τα τρία θεσμικά όργανα. Και έχω μεγάλες ελπίδες, καθότι εσείς είσαστε υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις, να καλέσουμε και τα τρία θεσμικά όργανα και να προκύψει ένα καλό αποτέλεσμα. Ε, Δεν βλέπω να έχουν ζητήσει άλλοι βουλευτές το λόγο. Α, ο Γουεντρέρο. Μισό λεπτό μόνο κύριε Πρόεδρε και κυρία Αντιπρόεδρε για να υπογραμμίσω την πολιτική σημασία που ενέχεται στα θέματα διαφάνειας. Τα τελευταία χρόνια στην πολιτική ζωή βλέπουμε ότι υπάρχουν πληροφορίες, αποκαλύψεις για συγκεκριμένες ε, συμπεριφορές οι οποίες πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Βλέπουμε τι έχει συμβεί σε διάφορα κοινοβούλια χωρών μελών ε, μη εξαιρουμένου του κοινοβουλίου της δικής μου χώρας. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι η διαφάνεια είναι καλύτερη από την απαγόρευση. Δηλαδή το να ε, υπάρχει ένας κατάλογος απαγορεύσεων χωρίς ε, ε, να αιτιολογούνται και χωρίς ε, και χωρίς κάποια στοιχεία συνοδευτικά κατά κανόνα οδηγεί σε παράβαση αυτών των απαγορεύσεων ενώ η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση είναι καλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι τούτο το βήμα είναι πολύ θετικό και συμφωνώ και με τους προλέντες συναδέλφους αλλά και με την Αντιπρόεδρο που είπε ότι θα πρέπει να είναι συνολικό το Μητρό και να εφαρμοστεί όχι μόνο για το Κοινοβούλιο την Κομισιόν αλλά για όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Εάν δεν υπάρχουν ε, άλλοι αγωνιτές θα ήθελα να δώσω... Α, κύριε Ντάφ και μετά ίσως να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριος Νταφ. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ξεκίνησα να λέω σχετικά με το δικό μας ε, εσωτερικό κανονισμό. Για να ενσωματωθεί καλύτερα αυτό το νέο μητρό ε, όπου θα καταγραφούν όλοι, όλες οι ομάδες πίεσης, λομπίστες κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνδυαστεί και με το πόθεν έσχεση, τις οικονομικές δηλώσεις των ε, μελών. και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να δείξουμε λιγότερη πειθαρχία ή λιγότερη αυστηρότητα. Και φρονώ λοιπόν πως ε, είναι μια ευκαιρία και για μας. Στα πλαίσια των αλλαγών του εσωτερικού κανονισμού να δούμε συνολικότερα τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ε, ο, ο κώδικας συμπεριφοράς για μας τους ίδιους τους βουλευτές. Και με τον τρόπο αυτό θα δείξουμε την σοβαρότητα με την οποία το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει το θέμα της ε, διαφάνειας Αυτά ήθελα να προσθέσω λοιπόν. Ωραία, να δώσουμε τώρα το λόγο ε, στον κύριο Κρίστιανσεν, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τη συζήτηση αυτή και εξ ονόματος του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων από πλευρά της Επιτροπής, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα που πετύχαμε. Είναι ένα τεράστιο βήμα προόδου προς την ε, κατεύθυνση της διαφάνειας για το πώς μας αντιλαμβάνεται ο κόσμος, πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τις εργασίες μας. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το μητρό πριν από τρία-τέσσερα χρόνια στα πλαίσια της διαφάνειας. Ήταν σαφές τότε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις διαδικασίες, υπήρχε πρόβλημα με την αντίληψη του κόσμου ως προς τις διαδικασίες. Άρα, ο μοναδικός τρόπος να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανησυχίες ήταν η διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν και ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία αυτή. Μας ικανοποιεί ε, το, η πρόοδος που έχει σημειωθεί και θυμάμαι όταν ξεκίνησα ε, πριν από 4-5 χρόνια ήταν ένας ε, μαγικός αριθμός. Ε, υπήρχε ένα σε όλες τις συζητήσεις. 15.000 ε, οργανώσεις αναφέρονταν ότι υπήρχαν. Κανείς δεν ήξερε αν ισχύει αυτό το στοιχείο, το αριθμητικό στοιχείο αυτό. Και όλοι τα αναφέραν λες και ήταν πραγματικό. Και τώρα να σας πω ότι έχουμε 3.500 καταχωρήσεις στην παρούσα φάση στο Μητρό μας και στο μέλλον θα έχουμε ένα κοινό μητρό και θα έχουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε μία ένδειξη, έναν ενδεικτικό ρυθμό των ατόμων που εργάζονται για τέτοιες οργανώσεις. Θα ξέρουμε ποιος είναι ε, ο υπεύθυνο του άτομο επαφής για κάθε οργάνωση και πώς λειτουργεί. Και ξέρουμε ότι τώρα έχουμε περίπου κάτι λιγότερο από 10.000 άτομα που καλύπτονται στο Μητρό. Είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν με την διαδικασία αυτή, αλλά να σας πούμε ότι πρόκειται για μια δυναμική ε, διαδικασία. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά σε 24 μήνες, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την διαδικασία αυτή. Δεν μπορούμε όμως να την ε, πιέσουμε, δεν μπορούμε τεχνητά να την επιταχύνουμε. Και όπως είπε ένας συναδελφός σας πριν από λίγο, υπάρχουν στοιχεία στο Μητρό το οποίο τα καθιστούν πιο υποχρεωτικό χωρίς να δίνουν ε, τυπικά υποχρεωτικό χαρακτήρα στην καταχώρηση στο Μητρό. Άρα μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πραγματευτούμε διάφορα στοιχεία για την αντιμετώπιση των όσων έχουν καταχωριστεί. Αλλά καλωσορίζω από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς το αποτέλεσμα και ε, συνεργαζόμαστε με τους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προετοιμάσουμε ε, μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι το κοινό αυτό μητρό προκειμένου να, προκειμένου να καταστεί λειτουργήσιμο προκειμένου να δείξουμε και προς τα έξω ότι υπάρχει μια λογική για το πώς συνεργαζόμαστε, πώς εργαζόμαστε στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα δώσω ξανά το λόγο στην κυρία Γουόλη, έτσι ώστε να απαντήσει στα σχόλια, στις ερωτήσεις κτλ. Εγώ ως ε, συνεισηγητής με μεγάλη προσοχή άκουσα όλα αυτά που είπε η κυρία Γουόλης και επομένως θα τα λάβω υπόψη μου. Κυρία Γουόλης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλια τα οποία κάνατε. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το ότι πολλοί συνάδελφοι έθιξαν το θέμα της διαφάνειας στο σύνολό της. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της νομοθετικής διαφάνειας. Και έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο ρόλο που μας έχει προδώσει η Νίκη της Λισαβόνας, ε, εκεί όπου ορίζεται ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερη διαφάνεια. Δεν ξέρω πώς από εσά έχετε συνειδητοποιήσει ότι είμαι η αντιπρόεδρος υπεύθυνη για τη διαφάνεια. Να η αρμοδιότητα μου στο Προεδρείο οπότε και κατά τη γνώμη μου που ε, είναι πάρα πολύ θετικό το να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτό το τομέα από κοινού, μια που τώρα θεωρώ ότι τώρα το κλίμα είναι πολύ πιο ευμενές, ε, υπάρχει πολιτική βούληση στο Κοινοβούλιο, είναι να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για αυτό το μητρό, αν θα είναι υποχρεωτικό ή όχι, ε, ε, στο γραφείο μου να σας πω τι κάνω. Αν έρθει κάποιος, και πει ότι ενδιαφέρεται, τον, τον ρωτάω, είσαι στο Μητρό. Και του λέω, εάν θέλεις να επανέλθεις μπορείς και προσοχή γιατί αν είσαι στο Μητρό μπορεί να μην είμαι και τόσο πρόθυμη. επομένω. θεωρώ ότι ε, όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να υπάρχει σε μια τέτοια μη υποχρεωτική μορφή ε, το Μητρό. τώρα έχουμε την ε, έκθεση αυτή του Φρίντριχ. Το Κοινοβούλιο το προώθησε και καλά έκανε, ούτως ώστε να υπάρχει κάποιο είδους νομοθετική απαρχή δημιουργίας τέτοιων εκθέσεων και είπαμε για όλα αυτά τα οποία έχουν επηρεάσει το γίγνεσθε οπότε και εμείς ως κοινοβούλιο θα μπορούσαμε νομίζω να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό τον του, του, του πόθεν έσχες γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τώρα θα διεκπληρωθούν ε, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο δυναμικά και επομένως και εγώ ως αντιπρόεδρος θα κάνω ό,τι μπορώ και θα προσπαθήσω να τα προωθήσω, να τα διεκπαιριώσω αυτά τα ζητήματα. Τώρα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά το Μητρό και όπως προείπαμε ε, προσπαθώ να σας τονίσω ότι με αυτή τη ε, ε, διαδικασία θέλουμε να υπάρχει υποχρεωτικότητα όσον αφορά αυτό το Μητρό και με μεγάλη μου χαρά να σας πω όποτε θέλετε τι, τι νομικές συμβουλές έχουμε λάβει από την νομική υπηρεσία Βέβαια ε, όπως ξέρετε πάντα οι, οι απόψεις των νομικών διήστανται αν θέλουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα ε, σε σχέση με τα όσα συμβουλεύει η νομική υπηρεσία και αυτό γίνεται. Πάντως τώρα είμαστε σε ε, άγνωστα ύδατα αλλά η συγκυρία είναι τέτοια που το κλίμα είναι ευμενές και από πλευρά συμβουλίου υπάρχει επομένω τώρα η ευκαιρία να κάνουμε βήματα προόδου και δεν θα ήθελα αυτή η ευμενής ε, συγκυρία τώρα να πάει χαμένη ε, υπάρχει επίσης και ο χρόνος ώστε Κοινοβούλιο και Επιτροπή από κοινού να προχωρήσουν προς ένα μητρό όπως ε, ε, προβλέπεται όπως τα είπαμε στις αρχές του θέρους αλλά τέλος πάντων ίσως τα πράγματα εξελιχθούν ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι θεωρούσαμε και τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνήσουν για την υποχρεωτικά του Μητρώου Βέβαια, κανείς μπορεί να ρίξει μια ματιά και στις νομικές συμβουλέ που έχουμε λάβει τώρα το θέμα του τι κάνουμε με τα φάουλ των ε, μελών των λόμπι. Κοιτάξτε τι γίνεται όσον αφορά τον κώδικα διοντολογία. Ε, ε, κάποιοι έχουν ενεργήσει αντιδιοντολογικά. Όμως όλα αυτά υπάρχουν στο Μητρό και υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις κυρώσεων σε σχέση με την άρνηση να τους επιτρέψουμε την προσβασιμότητα ανάλογα με το τι έχουν κάνει ε, φυσικά και μπορεί να γίνουν κάποιες έρευνες από τα θεσμικά όργανα και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος ενήργησε αντιδιοντολογικά, αντικανονικά τότε υπάρχει περίπτωση της δημόσιας καταγγελίας που είναι ίσως το πιο σημαντικό και πολύ εξημών θα θέλαμε να γίνει το εξή το οποίο γίνεται σε έναν βαθμό σήμερα. Εάν στις Βρυξέλλες οι εμπλεκόμενοι διαπιστώσουν ότι πρόκειται περί σοβαρού εγχειρήματο, τότε και αυτοί θα το πάρουν σοβαρά και θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δηλαδή, εάν είναι η λειτουργία του Μητρώου, τότε θα σκίζονται, ας το πούμε έτσι, οι λομπίστες να έχουν σαν παράσημο το ότι έχουν συμμετάσχει, είναι στο Μητρό, είναι άσπηλοι κλπ. κλπ. Επομένως είναι ένας ε, κύκλος, όχι φαύλος, αλλά ωφέλιμος επομένως. Διακόπτε. Ναι, ναι, ναι, υπάρχει το θέμα το λεπτό της Εκκλησίας. και δεν σας το λέω αυτά σαν ε, κλασικός φιλελεύθερος που είναι κατά της Εκκλησίας αλλά γιατί έχουμε το θέμα της πρωτοβουλία των πολιτών που έχει να κάνει και με αυτό το θέμα. Δηλαδή, εάν ε, έχουμε εδώ πέρα κάποιο επικάλυψη με αντίστοιχη πρόβλεψη για την Εκκλησία. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και αυτό το θέμα μας απασχόλησε αρκετά, λέει η κυρία Μας προβλημάτισε και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι, όπως και οι νομικοί, να έχουμε αυτούς τους εκπροσώπους της ε, Εκκλησίας και αυτοί Επίσης, ε, στο βαθμό που δραστηριοποιούνται στι Βρυξέλλε, και αυτοί να είναι καταχωρημένοι στο Μητρό. Βέβαια έχουμε αυτούς και έχουμε και κάποιους άλλους Τέλος πάντων, θα πρέπει όλοι να εγγραφούν στο Μητρό. Και όπω και οι νομικοί θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν αυτοί εμπλέκονται στην, στο πολιτικό γίγνεσθε, οπότε αναλόγω και εμείς θα κινηθούμε σε σχέση με το αν θα επιδιώξουμε αυτοί να καταχωρηθούν στο Μητρό. Άρα επομένω πρόκειται για τέτοιου ρύθμιση και δεν, δεν, δεν αποτελεί ε, βολή κατά τη εκκλησία. Πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το, ε, η συζήτησή μας. Υπενθυμίζω ότι το άρθρο 17 της ε, λειτουργίας της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, δηλαδή για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται σε έναν ανοιχτό και διάφανο ε, διάλογο και με τις εκκλησίες και τους εκπροσώπους της. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι επαφές, αλλά υπό το φως της ημέρας και όχι μυστικά και υπόγεια. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να καταγράφονται οι εκπρόσωποι των εκκλησιών εάν θέλουν να συζητούν μαζί μας. Εάν συμφωνείτε λοιπόν ε, να σας προτείνω το εξής χρονοδιάγραμμα. Μια και είμαι η εισηγητής για δύο εκθέσεις, μία για την έγκριση της ε, συμφωνίας για τη διαφάνεια και μια άλλη έκθεση η οποία θα αφορά τις ε, ε, κατάλληλες τροποποιήσεις κυρίως το άρθρο 9 του παραδείγματος 10 του κανονισμού προτείνω λέγω να έχουμε παρουσίαση των δύο προτάσεων στις 14 Μαρτίου έτσι ώστε η έγκριση να γίνει στη συνεδρία στις 19 Απριλίου και να περάσουμε στην Ολομέλεια τον Μάιο. Στην Ολομέλεια του Μαΐου λοιπόν να ολοκληρώσουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε νομίζω. Να ευχαριστήσουμε επομένω εκ βάθους καρδίας την Αντιπρόεδρο Wallis γιατί ήταν μαζί μας, αλλά βεβαίως και γιατί ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας ε, που ασχολήθηκε με το θέμα ε, γιατί λέω έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Το θέμα της ε, διαφάνειας είναι εξαιρετικά σημαντικό για το κοινοβούλιο μας. Σας ευχαριστούμε κυρία Γουόλης εκ βάθους καρδίας. Θα συζητήσουμε τώρα το σημείο 10, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η τροποποίηση λοιπόν του άρθρου 136 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με ένα μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Όμως ε, δεν έχουν φτάσει ακόμα οι εισηγητές. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα είναι εδώ μέχρι τις 10.30. Τώρα δεν ξέρω, θέλει κάποιο συνάδελφο να αναφέρει κάτι, να μιλήσει για κάποιο άλλο θέμα ή αλλιώ να διακόψουμε για πέντε λεπτά ή διαφορετικά να προχωρήσουμε στο σημείο 12, 13 και 14. Επόμενη ε, Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011, από τις 4 μέχρι τις 6 και μισή στις Βρυξέλλες θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση. Επίσης, μια άλλη έκτακτη συνεδρίαση, 17 Φεβρουαρίου 2011, από τις 10 μέχρι τις 12 στο Στρασβούργο και τέλος την κανονική μας συνεδρίαση, Δευτέρα 14 Μαρτίου, το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 6.30 στις Βρυξέλλες και 15 Μαρτίου η επόμενη μέρα, δηλαδή από τις 9 μέχρι τις 12.30 πάντα στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η τακτική μας συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά μας μένουν ακόμα πέντε λεπτάκια μέχρι τις 10 και μισή που θα έρθουν οι εισηγητές μας για το θέμα 10. Ε, θα διακόψουμε λοιπόν για 5 λεπτάκια, αλλά παρακαλώ να είστε όλοι εδώ 10 και μισή γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Allora, Allora, Πρόεδρος. Ξαναρχίζουμε λοιπόν την συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να εξετάσουμε το σημείο 10 της ημερησίας διατάξεως το οποίο είναι πολύ σημαντικό όπως σας είπαμε και πριν και αφορά την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με ένα μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη-μέλη του Eurogroup, ας πούμε, δηλαδή των κρατών που έχουν νόμισμα το ευρώ. Οι συγητές ε, από τις 27 Ιανουαρίου είναι οι Μπροκ και Γκουελτιέρη και εμείς θα πρέπει να εκφράσουμε την άποψή μας ε, σχετικά, ε, σύμφωνα μάλλον με την διαδικασία απλουστευμένης αναθεώρησης, άρθρο 138, και μετά από την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Φον Ρομπέι, ε, για την σχετική γνωμοδότηση από πλευράς μας. Δεν έχουμε χρόνο και επομένως θα πρέπει στη σημερινή συζήτηση να δώσουμε στους εισηγητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όλο το υλικό το οποίο θα χρειαστούν έτσι ώστε να εκπονήσουν την έκθεσή τους. Θα δώσω το λόγο στους ε, ε, δύο εισηγητές, δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος, ο κύριος Γουελτιέρη, ο κύριος Μπροκ. Ο ένας δείχνει τον άλλον. Τι να κάνω εγώ. Εντάξει, Γουελτιέρη λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση για ένα τόσο περίπλοκο και ευαίσθητο ζήτημα όπως αυτό της ε, τροποποίησης ε, της ε, συνθήκης της Λισαβόνας διαπλουστευμένης διαδικασίας έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ένα ζωτικό θέμα για την Ευρώπη, δηλαδή την δυνατότητα να έχει έναν σταθερό, έναν πάγιο μηχανισμό σταθερότητας πρέπει να πω ότι έχω πλήρη επίγνωση της εξαιρετικής ευαισθησίας του θέματος, καθώς επίσης και για, την, για το ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης που πρέπει να δείξει το Κοινοβούλιο. Όμως, πρέπει επίσης να πω ότι το να ασκεί κανείς με υπευθυνότητα το λειτουργήμά του θα πρέπει βεβαίως να γίνεται αλλά επί τη βάση της πραγματικότητας των αντικειμενικών δηλαδή και πραγματικών περιστατικών. Το αίσθημα ευθύνης δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει να δούμε και να αξιολογήσουμε σωστά αυτήν την πρόταση η οποία υπευλήθη από το Βέλγιο στην ουσία γιατί ο πρόεδρος του Συμβουλίου δεν έχει ε, δυνατότητα να υποβάλει μόνος του κάποιες προτάσεις. Με απασχολούν πολλά πράγματα. Είναι πολλοί οι προβληματισμοί μου που αφορούν και το θεσμικό σκέλος και τις πολιτικές επιπτώσεις αυτού του προεπιλεγέντος τρόπου δράσης αλλά και ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου που μας έχει υποβληθεί. Με συνθετικό τρόπο θα ε, σας πω τα στοιχεία που έχω και την επιχειρηματολογία μου για τα τρία αυτά θέματα. Πρώτον, αναθεώρηση λοιπόν του μηχανισμού με απλουστευμένη διαδικασία έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση αυτού του σταθερού, του μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας. Έχω πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι απαραίτητη από θεσμικής απόψεως μια τέτοια διαδικασία, για πολλούς λόγους. Διότι η νομισματική πολιτική των χωρών που έχουν το ευρώ είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαφώς καθορισμένη από το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία ενδεχόμενη ε, απόδοση στις ε, χώρες ε, μέλη για δυνατότητα αποκλειστικής νομοθέτησης, εάν αυτό συνέβαινε λέγω, ακόμα κι αν συνέβαινε θα μπορούσε να γίνει χωρίς τροποποίηση της συνθήκης. υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Εάν και εφόσον κάποιες χώρες απαιτήσουν ε, στην συνθήκη να γίνει συγκεκριμένη η αναφορά στη δημιουργία του μηχανισμού χωρίς την απλουστευμένη αναθεώρηση και αναφέρομαι εδώ στην δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρα ευελιξίας 352 ένα άρθρο το οποίο όμως θα πρέπει να αναγνωστεί ε, ε, ταυτόχρονα με την ετοιμιγορία του, του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας και που στην ουσία είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση. Σύμφωνα με την απόφαση αφενός ανεβαίνει πάρα πολύ το κατόφλι εφαρμογής της ρήτρας ε, ε, ευελιξίας βάσει της έννοιας competence competence και σύμφωνα με την απόφαση ε, όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 352 στην ουσία το δικαστήριο της Γερμανίας βάζει λίγο σε ίδιο επίπεδο και το άρθρο 352 και την ε, τροποποίηση. Και ε, λέει το δικαστήριο, χρειαζόμαστε εμείς, ας πούμε, στην ε, Γερμανία, ε, μία απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου έτσι ώστε να ξεκινήσει η μεταρρύθμιση, έτσι ώστε να αρχίσει η ισχύ της ρήτρας ευελιξίας. Ε, βεβαίως αυτή, αυτή η ρήτρα της ευελιξίας είναι πιο βαριά γιατί χρειάζεται πρώτερη ψηφοφορία κτλ. Πάντως προκύπτει εδώ εσωτερικό πολιτικό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς διαλέγουμε τη διαδικασία τροποποίησης της συνθήκης που απαιτεί 27 επικυρώσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο που με απασχολεί θέμα που παρουσιάζει, ενέχει πολλούς κινδύνους. Γιατί εάν πούμε ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργήσουμε το μηχανισμό σταθερότητας και γίνεται βάσει μιας πολύ απλής επιχειρηματολογίας που δεν μπορεί επομένως να τροποποιηθεί ε, με περαιτέρω απλούστευση το κοινοβούλιο ή ακόμα και ένα δικαστήριο όπως θα ήταν δυνατόν να γίνει στη Δανία μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή, τότε η Ευρώπη θα μπορούσε να βρεθεί ε, χωρίς καμία δυνατότητα ε, οικοδόμησης αυτού του μηχανισμού και επομένως οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πραγματικά δραματικές όσον αφορά την εξέλιξη του ενιαίου νομίσματος. Επομένως, είναι μεγάλη η ε, ευθύνη της επιλογής αυτού του μοναδικού εργαλείου και όχι κάποιου άλλου και δεν μπορεί να αποσιωπήσει τη σημασία του γεγονότος αυτού το κοινοβούλιο. Το τρίτο μου μέλημα, η τρίτη μου ανησυχία αφορά την ίδια την ουσία της επιχειρηματολογίας και του προτενόμενου άρθρου. Αφορά την τρίτη παράγραφο που προτείνεται στο άρθρο 136 και λεπτομερώς εξετάζοντας αυτήν την προσθήκη κατανοούμε ότι η επίπτωσή του σε πολιτικό και συνταγματικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Να δημιουργηθεί λοιπόν βάσει της τρίτης παραγράφου ένας μηχανισμός σε διακυβερνητική αποκλειστικά βάση και εντελώς απ' όχι μονάχα από την μέθοδο του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για ένα μηχανισμό που δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αφορά τα κράτη. Μα εάν αυτό ισχύει, τότε εάν δηλαδή τα κράτη μεταξύ τους δημιουργήσουν ένα μηχανισμό, τότε γιατί πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν χρειάζεται τροποποίηση των συνθήκων έτσι ώστε τα κράτη να κάνουν κάτι μεταξύ του γιατί εδώ μιλάμε για ένα μηχανισμό που θα βρίσκεται εκτός της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό με απασχολεί περισσότερο και θέλω να καταδείξω το γεγονός ότι η επιλογή να οικοδομήσουμε έναν μηχανισμό που θα είναι αποκλειστικά διακυβερνητικός μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις για την κατεύθυνση που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ας πούμε τους μηχανισμούς οικονομικής διακυβέρνησης. Εδώ γίνεται επιλογή τροχιάς, τροχιάς που όμως συνδέεται και με πολιτικές οθήσεις κατά κάποιο τρόπο που προκύπτουν από διαφορετικές ε, ιδέες ε, από κυβερνήσεις ε, που αντιτίθενται στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση αφενός ή από κράτη που θέλουν να δημιουργηθούν κάποιοι σκληροί πυρήνες πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καθαρά δηλαδή διακυβερνητική βάση. Αυτές οι δύο διαφορετικές πολιτικές οθήσεις μπορούν στην ουσία να ε, οδηγήσουν σε, έναν, σε μία οδό η οποία κινδυνεύει να μην είναι βήμα προς τα εμπρός. Κινδυνεύει να είναι οπισθοχώρηση, οπισθοδρόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα κείμενα που μας έστειλαν οι πολιτικές ομάδες ε, διαπιστώνω ότι υπάρχει και μία αντίκρουση ανάμεσα στην ε, ρεαλιστική αναγνώριση του γεγονότος ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αφενός και αφετέρου της άποψης ότι πρέπει να υπεραμεινθούμε μιας κοινοτική διαδικασίας. Δηλαδή θα πρέπει να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε αυτός ο μηχανισμός να λειτουργεί έτσι ή αλλιώς. Αλλά προσέξτε, εάν αποφασίσουμε να μπούμε στην οδό αυτή, τότε δεν θα μπορούμε πλέον να πούμε τίποτα για οτιδήποτε κάνουν κάποιες χώρες. Επομένως η επιλογή είναι βαριά, η επιλογή είναι πολύ ε, ε, σημαντική ενδεχομένως η Επιτροπή θα μπορούσε να κάνει κάποιες ας πούμε μη δεσμευτικέ, να διατυπώσει κάποιες μη δεσμευτικέ ε, προτάσεις αλλά δεν μπορεί να παρεμβαίνει πλέον. Εν πάση περιπτώσει αυτή η τροποποίηση θα μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τρόπο εάν πραγματικά πρέπει να γίνει ε, σημείο επί του οποίου εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες ακόμα. Η ιδέα μου θα ήταν μάλλον να ενταχθεί το άρθρο αυτό ε, σαν γράμμα γάμα ε, παύλα 1 ε, στο 136 που δεν θα άλλαζε τίποτε όσον αφορά το γεγονός ότι ομόφωνα οι χώρες του ευρώ θα αποφάσιζαν στα πλαίσια όμως μιας δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή στο Συμβούλιο στο Συμβούλιο, σε μια αίθουσα του Συμβουλίου και όχι σε μια άλλη αίθουσα στις Βρυξέλλες, την οποία θα έχουν κλείσει ε, για τη συζήτηση αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει έτσι ώστε ο μηχανισμός αυτός να συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επ' αυτού θα πρέπει η θέση του να είναι σαφής και ισχυρή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γουελτιέρη, λέει ο Πρόεδρος. Θα ακούσουμε τώρα τον δεύτερο εισηγητή, τον κύριο Μπροκ. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Να συμφωνήσω και εγώ με τις παρατηρήσεις του κ. Γκοτιέρη. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, δεν είμαι ακόμη σίγουρος για το πώς θα πρέπει να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Και γι' αυτό στις συζητήσεις αυτές εξαρτώμε και ο συνάδελφος Γκοτιέρη και εγώ μιλήσαμε και με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις γιατί αφενός έχουμε φυσικά κάποιες αντικειμενικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις και σε αυτό το σημείο συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκοτιέρη και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς στο τρέχον πολιτικό υπόβαθρο δεν θα αποτρέψουμε τα όσα πρέπει να γίνουν αλλά παράλληλα θα κάνουμε και αυτά τα οποία είναι εύλογα να συμβούν πέρα από τις δυνατότητες που ανέφερε ο συνάδελφος, δυνατότητα δηλαδή να πραγματευτούμε το άρθρο αυτό, μιλάμε για ένα κλασικό παράδειγμα ενισχυμένης συνεργασίας. Τα κράτη-μέλη με τη χρήση των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να συμφωνήσουν κάτι τέτοιο και αναφέρεται ανεκτά ότι μπορούν να συμμετέχουν όσοι πληρούν τους όρους και το καθεξής. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση ενισχυμένη συνεργασίας. Όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο θέλουμε να κάνουμε και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Η διακυβερνητική φάση είναι έντονη στη συγκεκριμένη φάση. Οπότε αυτός είναι ο λόγος και το αντικείμενο των εσωτερικών συζητήσεων και αυτός είναι ο λόγος που αναφέρεται ότι τα εθνικά κράτη ε, εγγυώνται τα χρήματα αυτά, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορεί να τα ε, εγγυηθεί. Και αυτό αποτελεί και το λόγο της δυσπιστίας προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που υπάρχει επί της αρχής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο πλευρές ίσως να ευθύνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει στα κρατημέλη ότι με τα μέτρα της είναι μη πολιτική και ότι δεν εμπλέκεται στις εσωτερικές συζητήσεις ε, ε, των κρατών. Και άρα δεν εμπλέκεται στην πολιτική πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα στοιχείο, Πρόεδρε, το οποίο θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε πέρα από το σημερινό σημείο τη ημερησία διάταξη. Είναι θέμα ιστορική οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσο όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους επιτρόπους και τον πρόεδρο της Επιτροπής κάθονται ε, στο κτίριο Μπερλεμόν, στα κτίρια τους, στα γραφεία τους. Γιατί είδαμε και στην περίπτωση πρώτη, αν δεν καταφέρουν να επιτελούν τα καθήκοντά τους ως υπουργεία, σαν να λέγαμε, και παράλληλα να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους Δηλαδή, όπως γίνεται και στις εθνικές κυβερνήσεις, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εθνική νομοθεσία, θα πρέπει ο εκάστοτε υπουργό να θεωρείται υπεύθυνο. Δεν μπορούμε να δρούμε ανεξάρτητα από την πραγματικότητα και αυτό λοιπόν μα έρχεται μπούμερανγκ με δραματικό τρόπο πλέον. Αυτό το σημείο θα πρέπει να το εξετάσουμε με καθαρό κεφάλι γιατί μας ε, φέρνει στην δύσκολη κατάσταση να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε τα καθοριστική σημασία μέτρα. Κοιτώντα το μηχανισμό κρίση και βλέπουμε και τι συζητιέται στι διάφορε κυβερνήσει, στι διάφορε πρωτεύουσε και στι Βρυξέλλε περί οικονομική διακυβέρνηση, ότι σκεφτόμαστε εκτό των πλαισίων τη συνθήκη. Μπορούμε να το αποτεχτούμε αυτό σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκη, αλλά σε μια τέτοια κατάσταση, αν οικοδομούμε μικρέ δομέ οι οποίε φαίνονται αθώες, τελικά θα καταλήξουμε με μεγάλες ε, δομές εκτός του πλαισίου του συνθήκων που θα είναι πέρα από τον έλεγχο των θεσμικών οργάνων. Γιατί πολύ απλά αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσει η όλη εξέλιξη και θα αποκαλυφθούν τα μας σημεία. Και φοβάμαι ότι είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής. Αν δεν προσέξουμε και αν δεν αντιληφθούμε το πρόβλημα που υπάρχει. Ότι υπάρχει πρόβλημα στα συγκεκριμένα σημεία. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αλλάξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κείμενο. Και δεν πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να να παίξουμε το παιχνίδι και να αποτρέψουμε αυτά που θα γίνουν στις 24-25 Μαρτίου. Γιατί η κατάσταση εκτακτών άγγιων των κρατών μελών και η επίδραση των ε, αγορών δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιτρέψουμε. Φοβάμαι ότι αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει και θα πρέπει να περάσουν τα όσα είναι απαραίτητα, ακόμα και αν είναι δυσάρεστα για κρατη Δεν θα λειτουργήσουν όλα με την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, αλλά αν υπάρχουν και δεσμεύσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση να ρυθμίσει τα ιστορικά της και να ληφθούν μέτρα που έχουν ληφθεί σε μια σειρά χωρών. Αυτό για τις ε, εθνικές κυβερνήσεις και για τα εθνικά κοινοβούλια είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο. Για μας είναι απλά τα πράγματα. Τα μέτρα λιτότητας δυσκολεύονται πάρα πολύ σε κάθε χώρα και αυτό ισχύει για όλους τους συναδέλφους από όλα τα κόμματα. Θα ληφθούν λοιπόν οι αποφάσεις 24 και 25 Μαρτίου. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα καταφέρουμε να έχουμε μια τοποθέτηση ωστόσο, τότε και να δούμε πώς θα προσπαθήσουμε, πώς θα επιχειρήσουμε να οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο την εφαρμογή προκειμένου να υπάρχουν σημεία ε, σύνδεσης για να εφαρμόζουμε αυτά που θέλουμε σε μετέπειτα ε, ε, ε, φάση. Για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάπτυξης είναι διακυβερνητικό. Το ΣΕΝΙΕΝ στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διακυβερνητικό και αυτό, εκτός των συνθήκων και ο τρίτος πυλώνας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, σε τελική ανάλυση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει το ρόλο, το ρόλο γραμματείας. Και νομίζω ότι πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε και πρόεδρο δεν είναι δυνατόν παρά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει πιο έντονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δημιουργηθούν νέες δομές όπως για παράδειγμα στην Ένωση για τη Μεσόγειο όταν είπαμε ότι, μας είπανε ότι θέλουμε το, η γραμματεία της Ένωσης και τη Μεσόγειο στο Παρίσι και παρόμοια, πολλά τέτοια παρόμοια παραδείγματα. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να θέσουμε ένα ορόσημο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε πλειοψηφία μέχρι 24-25 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους ε, αναφερόμενους λόγους αλλά θα πρέπει να υπάρχει προθυμία από το Συμβούλιο και θα πρέπει να υπάρχει και θέληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι προς το συμφέρον τους, που θα μας δώσει τη δυνατότητα αυτός ο διακυβερνητικός τομέας αποφάσεων να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να μπορέσει εν καιρό να ενταχθεί στην κοινωτική πολιτική και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μας στοιχείο, νομίζω το πρώτο σημείο αναφοράς. Και εδώ θεωρώ ότι υπάρχει και μία αίρεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κινηθούν τα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν προτείνει ο συνάδελφος Γκοτχέρη, πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με όλες τις προτάσεις. Είναι πάρα πολύ καλές, πολύ καλύτερες από τις δικές μας. Από τις δικές μου. Τι από αυτά όμως είναι εφαρμοστέο. Και κατά δεύτερον, θα πρέπει στην έκθεση, στην έκθεσή μας να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε ευρέως την κατάσταση, να ε, ε, ε, περιγράψουμε επακριβώς τη συνολική κατάσταση και από τις διάφορες επιτροπές παρουσιάζει ο καθένας τη δική του θέση. Πρόκειται για μια συνολική λοιπόν αντίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο, στην έκθεσή μας. Να συμπεριληφθεί το θεσμικό πλαίσιο και να διευκρινίσουμε την πολιτική σημασία. Πιστεύω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να έχουμε και μία μικρή επιρροή προκειμένου να θέσουμε τους όρους για τις μελλοντικέ εξελίξεις. Και θα ήθελα να ακούσω πώς ε, τα αντιλαμβάνεστε εσείς κύριε Πρόεδρε και πώς τα αντιλαμβάνονται και οι συνάδελφοι και έτσι να τα συμπεριλάβουμε και τις δικές σας προτάσεις μαζί με τον κύριο Κοτιέρη και να τις υποβάλουμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Μας τα προβλήματα που είναι σοβαρά και Είδαμε επομένως τη διάσταση του θέματος και έχει ζητήσει το λόγο πρώτος ο κύριος Νταφ. Uh, the... Κύριε Πρόεδρε, η πρόκληση είναι να έχουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας, ο οποίος δεν θα αντιβαίνει ή στο άρθρο 125 της συνθήκης σε σχέση με τις διατάξεις για οικονομική ενίσχυση και σωτηρία ούτε θα ακυρώνει ε, την επιταγή για τέλεση δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ 100% ευθυγραμμίζομαι με τις ε, επιφυλάξεις εκείνες που αφορούν τον διακυβερνητικό χαρακτήρα αυτού του μηχανισμού σταθερότητας εκείνες που διατυπώθηκαν από τον Έλμαρ Μπρόκ και τον Γκουαλτιέρη. Προτιμότερο είναι Εάν δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, σαν ενωσιακό τμήμα του συστήματος, τότε να θεωρήσουμε ότι αυτό το οποίο θα φτιάξουμε τελικά θα ενταχθεί στο ενωσιακό σύστημα, ακριβώς όπως έγινε και με το Σέγγεν και με επιτυχία. Όμως, έχουμε και το παράδειγμα το οποίο είπε ο κύριος Μπρόκ που δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και την ε, Μεσογειακή Ένωση, διότι καμία από αυτές τις δύο προσπάθειες δεν ακολούθησαν αυτή την ε, πορεία την οποία θέλουμε τώρα να ακολουθήσουμε. Άρα και πρέπει κανείς να αντλήσει τα αντίστοιχα συμπεράσματα από αυτές τις ατυχείς εμπειρίες του παρελθόντος. Οπότε και δεν διαμορφώθηκε συνένεση στα πλαίσια της συνθήκης και επομένως ακολουθήθηκε μέθοδος εκτός συνθήκης. Όπως είπε ο εισηγητής, έχουμε το άρθρο 352 σαν εναλλακτική λύση που προβλέπεται από τη συνθήκη. Βέβαια προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι μια εναλλακτική λύση τόσο ελκυστική από πλευρά νομική. Επίσης, εδώ συντρέχει το άρθρο 329 κατεξοχήν νομική βάση για την ε, ενισχυμένη συνεργασία. Επίσης έχουμε και το άρθρο 133. Το άρθρο το οποίο προβλέπει για τα αναγκαία μέτρα αναγκαία για την χρήση του ευρώ. Και οπότε πριν καταλήξουμε σε μια άποψη ως κοινοβούλιο να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να κάτσουμε και να διερευνήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις. Επίσης, όπως είπε και ο κ. Μπρόκ, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, ούτως ώστε να δούμε πώς θα θέλαμε να έχουμε μια αξιόπιστη οικονομική διακυβέρνηση. Κάτι το οποίο αποκλείεται να προκύψει από το Συμβούλιο και φοβάμαι ούτε από την Κομισιόν. Κατά τη γνώμη μου, μάλλον απορτουνιστικά ενεργή για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά θα πρέπει κανείς να σκεφτεί στρατηγικά, να αποφασίσει πού θέλει να καταλήξει αυτή η προσπάθεια, μια που αυτή θα μπορούσε να είναι μόνο η πρώτη από μια σειρά αλλαγών. Και όπως είπε ο κύριος Μπροκ, θέλουμε να έχουμε τελικά μία εκβάθρον αναδιοργάνωση της ε, Επιτροπής και να φτάσουμε σε μέτρο βαθμό αυτοματισμών όσον αφορά την επιβολή κάποιων κυρώσεων για τις οποίες προϋποτίθεται μια τροποποίηση του άρθρου 124 Κάτι που έχει σχέση και με την εκπροσώπηση του Eurogroup και επίσης χρειάζεται και να υπάρξει κάποιος ταμιακή ευκολία από πλευρά τη Επιτροπή, δηλαδή να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα, στην οποία να έχει προσβασιμότητα η Κομισιόν, αλλά επίση και συντονισμό και συνεργασία με το Eurogroup τη Κομισιόν και να έχουμε κάποιο είδου γνωμοδότηση, ψήφισμα, όπου θα πρέπει να διατυπώνουμε ε, τις πιο μακρόπνοες επιθυμίες μας για μια αξιόπιστη οικονομική διακυβέρνηση. Επίσης, κατά τέτοιο λόγο, θα πρέπει να ε, επιμείνουμε και να ενισχύσουμε την θέση του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ε, μεταρρύθμιση του όλου συστήματος ιδιών πόρων. Η πολιτική μας ομάδα άρχεται πάρα πολύ στις ε, απόψεις του κυρίου Λαμασούρ. Και όλοι θα πρέπει τελικά να εμπλακούν και τεχνικά εθνικά κοινοβουλία για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, προοπτικέ που υπάρχουν για την ε, στήριξη του ευρώ. Άρα, μέσα σε ένα θα πρέπει όλα αυτά να τα προτάξουμε ως απόψη του Κοινοβουλίου και θα ήταν πάρα πολύ θετικό το έργο μας. Επίσης, εάν μπορούσαμε να έχουμε επαφές με Ρεν και Τρισέ, γιατί οι τρεις καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε και άρα θα πρέπει να έχουν κάποια συνέπεια συνοχή οι απόψεις μας. Μην έχουμε απόκληση των απόψεών μας. Γιατί σε τέτοια περίπτωση φυσικά αυτό θα έχει μοιραία αντίκτυπο στις αγορές. Άρα θα πρέπει και η Κομισιόν, ο Επίτροπος και ο κύριος Τρισέ να μας πούν μας πούνε ακριβώ, τι, τι γίνεται, πώς λειτουργεί, πώ ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός σταθερότητα ευρωπαϊκό. Να μα πούν επίσημα, δημοσία, τις ε, απόψεις Αλλά και ποιο θα είναι το κόστος κάποιου δανείου διευκόλυνσης διάσωση για το κράτο το οποίο ενδεχομένω πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Τέλος, θα ήθελα οι συνάδελφοι τι πρεσβεύουν, γιατί κατά τη μου πρόκειται για ένα περίπλοκο, για ένα δύσκολο θέμα, οπότε και θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες μας. Προσωπικά θα προτιμούσα στη δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου δηλαδή στις 24 του μηνός, την 5η, τότε να ψηφίσουμε ακριβώς πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οπότε και ο πρόεδρος Μπούζεκ θα μπορούσε με το κείμενό μας την γνωμοδότηση να πάει έτσι εις το Συμβούλιο και κατά αυτόν τον τρόπο θα τονιζόταν περισσότερο η κρισιμότητα, σοβαρότητα με την οποία το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Μέντες Δεβίγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους συζητητές για αυτή την πρώτη εισαγωγική, προσαγωγική συνεδρίαση για την ε, πρόταση του Συμβουλίου όσον αφορά την ε, τροποποίηση του άρθρου 136. Για να δούμε τι ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Ζητάμε δύο πράγματα. Να μας πούν πρώτα-πρώτα, εάν συμφωνούν, να γίνει μια διακυβερνητική διάσκεψη. Να μας πούν ναι ή όχι. Για ποιο λόγο να γίνει, ούτω ώστε έτσι να τροποποιηθεί το άρθρο 136, ακριβώς όπως αποφάσισε το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμένα μου φαίνεται σωστή αυτή η διαδικασία. Το άρθρο 48. Το 308. Está para, para Παλιό 308 Είπαμε ότι είναι πρόσφορη νομική βάση, όμως είδαμε πόσο αυτό είχε προβληματίσει τα κράτη-μέλη γιατί προϋπέθεται ή τέλος πάντων επέφερε κάποια μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα κράτη-μέλη στην Ένωση. Άρα το 352 συγκροτεί έναν ολόκληρο μηχανισμό που μπορεί να επιφέρει ε, κάποιες ε, πρωτοβουλίες από μόνο του δεν είναι μηχανισμός δημιουργεί επομένως είπαμε ότι με την σημαίνει συνεργασία και το 133 και το ευρώ κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε κάτι σαν εμβριουλικό έχουμε κάπως κάτι σαν ε, ζορισμένη λύση και ερμηνεία επομένως κατά τα άλλα εντάξει οπότε γι' αυτό και όπως σας είπα θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πει αν συμφωνεί ή όχι με μια τέτοια διάσκεψη και μια που σήμερα ε, έχουμε αυτή την ε, κρίση που μας ε, μαστίζει όταν το Συμβούλιο θέλει να στείλει ένα μήνυμα σταθερότητας στις αγορές τότε νομίζω ότι θα ήταν λάθος το Κοινοβούλιο να αρχίσει να έχει αμφιβολίες, ε, ενστάσεις για αυτή την, ε, ε, για αυτή την διαδικασία και να αρχίζει να βάζει τροχοπέδες σε αυτό το μηχανισμό. Θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε ασφάλεια και οι θεωρητικές συζητήσεις για τις εναλλακτικέ λύσεις σωστές είναι, όμως θα πρέπει να ολοκληρωθούν πάρα πολύ σύντομα και να βιωτώσουν προσοχή μας στο πιο ουσιώδες. Αυτή είναι η γνώμη μου όσον αφορά αυτές τις ε, αμφιβολίες για τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα την ουσία, Πρόεδρε, το Συμβούλιο διατύπωσε μια συγκεκριμένη πρόταση και θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να γίνει μια τροποποίηση αυτής. Προβλέπετε και νομικά. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια τέτοια αναθεώρηση τροποποίηση. Οπότε Αυτό το λένε και οι εισηγητές. Καλός, κακός, αυτό το προτείνουν. Επομένως, κινούμαστε σε αυτό το πλαίσιο σήμερα. Και θεωρώ ότι αυτός ο μόνιμος μηχανισμός είναι ένα εργαλείο, ένα κομμάτι ενός μηχανισμού. Πρόκειται για κάτι που πρέπει να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά και αν μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί αυτή η ψηφίδα θα μπορεί να μπει στο όλο μοσαϊκό ε, οπότε μετά το σύνολο του μοσαϊκού θα βοηθούσε στην οικονομική διακυβέρνηση και επομένως είπαμε ότι προσέχουμε πιο πολύ την νομισματική παρά την οικονομική ένωση τα έχουμε πει αυτά και ε, όσον αφορά εκείνη την ε, διάσκεψη που προετοίμασε το Σύνταγμα και ε, το στο έργο που επετέλεσε ο φίλος Κλάους Χένς, τελικά δεν καταλήξαμε σε καμία απόφαση γιατί τότε θεωρούσαμε ότι δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν εκείνες οι διατάξεις που είχαν θεσπιστεί στην νίκη του Μάστιγκ Τώρα όμως άλλαξαν τα πράγματα και καταλάβαμε ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή και σε αυτό το μέτωπο. Επομένως τώρα υπάρχει το θέμα της κοινή γνώμη, όπω είπε ο πρόεδρο Καζίνη θέμα επικοινωνιακό δηλαδή και να δούμε κατά πόσον θα φανούμε ικανοί να, να παραδεχτούμε, να προτάξουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά την Οικονομική Ένωση. Είναι επομένω τώρα μια μοναδική ευκαιρία που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσει να εξηγήσει στην κοινή γνώμη, στα πλαίσια αυτού του, του μοσαϊκού, αυτού του, του, της ψηφίδας, που θέλουμε να βάλουμε στο μοσαϊκό για το ποια θα είναι η συνολική εικόνα. Οπότε, ετήσι των Γκολτιέρη και Μπρόκ, οι συντονιστές, κάτσαμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κείμενο όσον αφορά τον πολιτικό παιδαγωγικό μας ρόλο, το δηλαδή το πώς θα δείξουμε το πώς θέλουμε όλα αυτές οι ψηφίδες να ενταχθούν σε αυτό το μοσαϊκό. αυτή η έξι κανονισμοί που αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση. Συνολικά και πώς όλα αυτά θα συνδέονται στην πολιτική για την Ευρώπη του 2020 αλλά και όπως είπε ο κύριος Νταφ στο τι θα γίνει με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα μπορέσουμε και πώς θα μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά τα οποία τώρα βρίσκονται επί της τραπέζης και να σας δώσω ένα παράδειγμα για το τι θέλω να πω. Να πάμε παραπέρα δηλαδή από τις προτάσεις της Κομισιόν όσον αφορά τα παραστρατήματα των κρατών μελών γιατί αυτά τώρα είναι λόγια, μπλα μπλα. Ε, επομένως, δεν θα πρέπει να μένει κανείς σε κάποια σύσταση δεν θα πρέπει να, να είναι κάτι σχεδόν σαν χάρτη σε, στα κράτη που δεν πάνε καλά. Θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω αυτό το οποίο κάνει η Ευρώπη. Και επομένω, να δούμε πώ όλα αυτά θα συντεριάξουν και πώ θα στείλουμε το μήνυμα τη ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη σοβαρότητα, γιατί αυτό ζητάει η Ευρώπη σήμερα. Και γι' αυτό και εγώ επιμένω. Νομίζω ότι θα πρέπει ξεκάθαρα να απαντήσουμε σε αυτό το οποίο μας ρωτάνε για αυτή τη διαβούλευση. Δεύτερον, θα πρέπει να ε, εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και στην εν λόγω έκθεση να μπορέσουμε να περιλάβουμε αυτή την συνολική εικόνα για το πώς θα πρέπει να έχει, πώς θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση και επίσης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με το, το, το, χρονικό πλαίσιο. Να είμαστε πιο περιοτικοί και να μην βυζαντινολογούμε. Ξέρω ότι δουλεύουν σκληρά οι συγητές. Πολύ καλό το ότι έχουν επαφή και με το Φανερομπάι. Και άρα επομένως πριν τη Δευτέρα, γιατί, γιατί ο χρόνος πιέζει, πριν τη Δευτέρα να έχουμε μία έκθεση που να εξετάσουμε, γιατί τελικά με την έκθεση αυτή θα πρέπει από το Κοινοβούλιο να πει ένα ναι ή ένα όχι σε αυτό που του ζητούν, το κατά πόσο θα γίνει όχι μία διακυβερνητική. Και φυσικά εγώ λέω ότι ναι, να πούμε ναι, ε, όπως βλέπει το 48-6 να προχωρήσουμε προς διακυβερνητική χωρίς πολλά πολλά. Και επομένως έχουμε αυτό το χρονικό πλαίσιο και αυτό χρειάζεται τώρα η Ευρώπη, σταθερότητα, ασφάλεια και επομένως να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Ναι, να και έχουμε και έκτακτες συναντήσεις όπως είπε ο κύριος ε, Ντάφνα, να φωνάξουν τον Τρισέ, τον Ρέν κλπ. Αλλά το χρονοδιάγραμμα να μην τεθεί ένα αμφιβόλο γιατί τότε αυτό θα είναι το λάθος πολιτικό μήνυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους άλλους μιλητές, θα ήθελα να πω ότι εγώ θα ήθελα κάποιες αποσαφηνήσεις. Ο συνάδελφος μιλάει για την ε, σύγκληση της ε, ε, διάσκεψης. Ναι, αλλά το Συμβούλιο ζητάει απλουστευμένη διαδικασία, συνάδελφε Μέντες Δεβίγο. Δεύτερο ερώτημα. Απάντηση εκτός μικροφώνου δεν ακούνε διερμηνείς. Τα ισπανικά μου είναι πολύ κακά. Εγώ είπα ότι είμαι υπέρ της διαδικασία 136 βάσει τη αποστολής διαδικασίας. Καμία αμφιβολία επ' αυτού. μάλλον κατάλαβα λάθος. Εντάξει, επομένως το θέμα σας είναι σαφές. Δεύτερον, να ρωτήσω τον κύριο Γκουελτιέρη ε, μια μεγαλύτερη αποσαφήνιση σχετικά με τα θετικά στοιχεία τα οποία τα οποία θα προέκυπταν από το ε, εάν το σημείο εγγράφεται ως γάμα στο 136 ή ως ε, παύλα στην παράγραφο 3 του 136. Μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά. Ο συνάδελφος Μάρτιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι μετά από αυτά που είπε ο Μέντες Δεβίγο είναι πιο απλή η παρέμβασή μου γιατί συμφωνώ απολύτως με όσα είπε. Είμαι υπέρ της απλουστευμένης διαδικασίας και υπέρ της προτάσεως του Συμβουλίου. Συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συζητούμε τροπολογίες ε, Ε, μιλάμε για δημοσιονομικά και έχουμε την αίσθηση ότι αν δεν κάνουμε κάτι ε, τότε θα πέσει ο κόσμος αλλά εννέα στις 10 φορές αυτό δεν ισχύει. Εδώ μιλάμε ε, όμως για ένα πράγμα επί του οποίου αν δεν έχουμε ε, θετική αντιμετώπιση τότε πραγματικά θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι μονάχα σε απλές ε, ταραχές των αγορών και διακυμάνσεις των αγορών αλλά μιλάμε για χώρες οι οποίες θα πτωχεύσουν και επομένως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ο Ρομπέρτο μίλησε πολύ ε, ε, πολύ ενεργητικά κατά της πρότασης και μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που λέει αλλά εδώ πρέπει να δράσουμε γιατί έχουμε απέναντί μας τον πραγματικό κόσμο και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τον πραγματικό κόσμο. Βεβαίως βλέποντας την πρόταση μπορούμε να πούμε ότι ε, προσπαθεί να βάλει το Συμβούλιο μια διακυβερνητική η οποία θα στενέψει πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι μια σέλα πάνω από, το κοινοβούλιο, πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να συμφωνήσω, αλλά από την άλλη πλευρά ε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι θα ενταχθεί σιγά σιγά στο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να γίνει αυτό μέσω τροποποίησης τη νομικής βάσης στην ε, πράξη, ε, στην χρήση αυτού του μηχανισμού σταθερότητας που προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι κι αλλιώς θα πρέπει ενεργότατα να συμμετάσχει οι κυβερνήσεις δεν θα έχουν μια διακυβερνητική γραμματεία. Επομένως οι προτάσεις ε, ε, σχετικά με την άσκηση του μηχανισμού σταθερότητος, ε, αυτός που θα ελέγχει, αυτός που θα επιβλέπει, αυτός που θα επιβάλλει, σίγουρα θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός που θα έχει τις σχέσεις με, το, με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομιζωτικό Ταμείο θα είναι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα ενταχθεί στην δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και εγώ δεν βλέπω τη διαδικασία σαν απλουστευμένη διαδικασία, αλλά σαν ένα απλουστευμένο ναι. Πρόκειται για ε, ε, μια, μια στιγμή μεγάλης έντασης στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίως μπορούμε να βάλουμε αιρεσιμότητες στην πρότασή μας ε, και θα υπάρξουν κοινοβούλια όπως ας πούμε σίγουρα το Βρετανικό Κοινοβούλιο που θα πούν κοιτάξτε όχι αυτή η πρόταση ξεπερνάει αυτά που μας είχατε πει αρχικά άρα δεν συμφωνούμε, απορρίπτουμε την πρόταση. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση όσο γίνεται απλούστερο και γρηγορότερο ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο μονάχα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς ένα πιο αποτελεσματικό και εν πάση περιπτώσει λειτουργικό νομισματικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρο. Ο Μάρτιν είπε ότι ο Μέντες Δεβίγκο έκανε πιο απλή την εισήγησή του. Ε, ο κύριος Μάρτιν έκανε τη δική μου εισήγηση ακόμα πιο εύκολη. Σύμφωνα απόλυτα. Με την προπτική την οποία παρουσίασε ο συνάδελφος Μέντες Δεβίγκο. Και με τον τρόπο που παρουσίασε, θα έλεγα, την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις θεσμικές σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί ο Ντέβεντ Μάρτιν ε, παρουσίασε με σωστό τρόπο τις δυναμικές αυτές σχέσεις. Θεωρώ ότι έχουμε κάθε λόγο να τονίσουμε στο σημείο αυτό μία από τις δύο ιδέες τις οποίες ε, παρουσίασε ο Ρομπέρτο Γκοτιέρη. Καταρχάς, την ευθύνη και κατά δεύτερον, το νομικό επιχείρημα και την κοινοβουλευτική θεώρηση, την παραδοσιακή θεώρηση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Σε θέματα, ωστόσο η υπευθυνότητα, η ευθύνη θα πρέπει να είναι πιο υπογραμμισμένη στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω, μάλλον δεν θα ήθελα να παρουσιάσω τα νομικά επιχειρήματα, τα παρουσιάστηκαν άλλωστε πάρα πολύ ορθά από τους δύο προλαλήσαντες. Από τον κύριο Μέντες Δεβίκο και από τον Μάρτιν. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει και ένα πολιτικό επιχείρημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δεν είμαστε νομικοί λέσχοι. Ξέρετε, είμαστε πολιτικοί. Ασκούμε πολιτική κάθε μέρα. Και έχουμε ένα θεσμικό, πολιτικό ζήτημα, πρόβλημα να επιλύσουμε. Θα πρέπει λοιπόν με πολιτικό τρόπο, πολιτικό πώ να ανταποκριθούμε και να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω απόλυτα τι θέσει των συναδέλφων, των δύο συναδέλφων, γιατί πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει σκοπός στο σημείο αυτό. Αν δεν αντιληφθούμε τι συμβαίνει σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, ίσως και την Ισπανία κατά πάσα πιθανότητα. Και πώς άλλες χώρες που βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση, ιδιαίτερα οι εθνικοί βουλευτές, πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Mm. Πώς αντιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και οι Γερμανοί την κατάσταση Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Και με όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν υπόψη, θα πρέπει να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση υπέρ του μηχανισμού αυτού. Και της απλής επίλυσης του προβλήματος, της όσο πιο απλής επίλυσης γίνεται. Αυτή της άποψη είμαι. Ασφαλώς, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε ότι ο μηχανισμός αποτελεί ένα μόνο στοιχείο μια συνολικής ανταπόκρισης, πρέπει να τα πράξουμε. Και όπως είπε ο Έλμαρ Μπροκ, κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να δώσουμε και το συνολικό υπόβαθρο στην έκθεση αυτή, το συνολικό υπόβαθρο της απόκρισής μας. Αν μπορούμε ασφαλώς να κάνουμε κάτι για να εμπλέξουμε πιο επίσημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό πάντα είναι ε, προς όφελος της διαθεσμικής ισορροπίας και του Κοινοβουλίου. Γιατί υπό την ιδιότητά μας ως ελεγκτή και συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είμαστε πιο ισχυροί παρά υπό την ιδιότητά μας να, ε, στις επαφές μας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ασφαλώς, αν μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το επιδιώξουμε. Αλλά στη τελική ανάλυση πρέπει να τονίσουμε, θεωρώ, τον στρατηγικό σκοπό, το στόχο της πολιτικής μας ευθύνη. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη, αλλά και σε συνάρτηση με τα άλλα θεσμικά όργανα, θα είναι σε καλύτερη θέση αν επιδείξει μια ρεαλιστική και υπεύθυνη στάση παρά αν υπερασπιστεί και προασπιστεί ένα θεωρητικό όραμα της θεσμικής μας θέσης. Στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου, του διαθεσμικού πλαισίου. Αυτό είναι το πολιτικό επιχείρημα που θα ήθελα να εισέλθει στη συζήτηση. Όχι τώρα αν πρόκειται για το άρθρο 352, 355 κτλ. Θεωρώ ότι αυτά μπορούν να γίνουν εύκολα αν γνωρίζουμε από πολιτική σκοπιά, από στρατηγική σκοπιά τι θέλουμε να πετύχουμε στην παρούσα φάση. Έφνερ. Yeah, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο εισηγητές. Γιατί θεωρώ ότι με πολύ καθαρό τρόπο παρουσίασαν το πρόβλημα και αυτό θεωρώ ότι είναι το καθήκον της Επιτροπής μας, όχι ε, γρήγορα και πρόχειρα να επεξεργαζόμαστε τα όσα μας αναλογούν, αλλά να παρουσιάσουμε με καθαρό τρόπο το πρόβλημα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θεσμικές συνέπειες και Συνάδελφε, αυτό το... Συνάδελφε αυτό δεν το κάνουμε για θεωρητικούς λόγους σήμερα, όχι, αλλά επειδή μας έχουν εκλέξει για αυτόν τον σκοπό οι Ευρωπαίοι πολίτες και έχουμε καθήκον να φροντίσουμε η Ευρώπη να τηρεί τους κανόνες που η ίδια έχει θέσει. Θα πρέπει να πω ότι όπως ε, πολλοί συνάδελφοι δεν έχω καταλήξει σε μια οριστική άποψη, σε μια οριστική τοποθέτηση. Αλλά στη σημερινή συζήτηση θα ήθελα να πω με πάσα σαφήνεια ότι η απλοποιημένη διαδικασία τραποποίησης της συνθήκης, την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, θεωρώ ότι αποτελεί μια λύση για επουσιώδεις αλλαγές της συνθήκης. Δεν αποτελεί μια εναλλακτική διαδικασία σε ό,τι αφορά μεγάλες και σημαντικές αλλαγές της συνθήκης. Αυτό που επί της παρούσης συζητάμε, η ασπίδα διάσωσης, αποτελεί ένα μόνο στοιχείο ενός συνολικού προβλήματος. Αυτό που με ανησυχεί επί του παρόντος λοιπόν είναι ότι μιλάμε και περνάμε αγκομαχώντας από ένα μικρό μέτρο σε ένα άλλο μικρό μέτρο και χάνουμε ίσως το σύνολο θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο θεσμικό πρόβλημα. Και ποιο είναι αυτό, το ότι αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο, αυτά που συνέβαιναν και ρυθμίζονταν καλώς ή κακώς ε, σε επίπεδο κράτους μέλους παλαιά, παλαιότερα, για το πώς εγγυόμαστε, για παράδειγμα, τα χρήματα σε έναν ισολογισμό πλέον καταδεικνύει ότι δεν έχουμε δημιουργήσει τα ε, σωστά όργανα, τα σωστά πλαίσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε και ένα θέμα με τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης και το πώς αυτά σχετίζονται με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να επιλύσουμε τα θέματα αυτά. Ιδάλλως διαρκώς θα ανακύπτουν προβλήματα τα οποία δεν θα μπορούμε διαρκώς να επιλύουμε με ασπίδες διάσωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι υφίσταται ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι πολλές, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει οικονομικές συνέπειες αλλά και θεσμικές συνέπειες. Ανακύπτουν θεσμικά ερωτήματα. Ιδιαίτερα από πλευράς θεσμικής λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτούμε. Χρειαζόμαστε κάποιες διαδικασίε για την δημοκρατική νομιμοποίηση και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι είναι επιτακτικό το καθήκον να τα δούμε όλα αυτά σε συνάρτηση το ένα με το άλλο και θεωρώ ότι είναι καθήκον και της Επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και συμφωνώ με τις ανησυχίες που εξέφρασε ο συνάδελφος Κοτιέρη και ο συνάδελφος Μπροκ ότι όλο και πιο πολύ στην παρούσα φάση προσπαθούμε να επιλύσουμε τα θέματα διακυβερνητικά το οποίο ουσιαστικά για θέματα τα οποία ουσιαστικά θα βρουν βιώσιμη λύση μόνο σε κοινωτικό επίπεδο και να μην ε, απατώμαστε διακυβερνητικό επίπεδο τι σημαίνει ότι είναι πολύ περιορισμένες οι κυβερνήσεις οι οποίες ε, συμφωνούν για έναν τρόπο, μια κατεύθυνση χαράσουν μια πολιτική η οποία γίνεται τελικά πολιτική της Ένωσης αλλά δεν γίνεται τελικά η συζήτηση για το τι θα είναι πιο ωφέλιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν ανησυχώ ιδιαίτερα και θα ανησυχούσα, θα ανησυχούσα ιδιαίτερα αν συμφωνούσαμε ε, χωρίς ε, οποιαδήποτε όρο στην απλουστευμένη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε εγγύηση ότι τα επόμενα βήματα θα γίνουν με άλλη διαδικασία. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα ακολουθείται διαρκώς αυτή η οδός και διαρκώς θα συμφωνούμε σε τροποποιήσεις στις συνθήκες και ότι θα μας παρουσιάζονται συνεχώς ε, τροποποιήσεις για τις οποίες θα μας λένε ότι θα πρέπει να περάσουν γρήγορα-γρήγορα». Είμαι λοιπόν επί της αρχής κατά της χρήσης ε, αυτής. Αν είχα την εγγύηση ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, πιο εύκολα θα συμφωνούσα στην προτινόμενη τροποποίηση. Και συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτό που είπε ο Άνδριου Νταφ. Να μην βιαστούμε και τα απασαλείψουμε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το, την όλη διαδικασία θα πρέπει να επιμείνουμε στη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και τελικά να ψηφίσουμε τέλη Μαρτίου στην Ολομέλεια. Ευχαριστούμε. Γιώργο Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε το λόγο. Ελπίζω δεν θα ακρηγορήσω και θα είμαι όσο γίνεται απλός γιατί θεωρώ ότι οι πανεβάσεις των συναντήλων που έχουμε σήμερα όλες μας οδηγούν στο ότι ως συμπέρασμα και στο παρελθόν όπως έγινε και σήμερα το Κοινοβούλιο περισσότερο από όλους αντιπροσωπεύει το όραμα το ευρωπαϊκό. Οικονομικό, νομισματικό και κυρίως πολιτικό και ο κύριος Μπροκ μας ανέφερε ότι στον 13ο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκεί ψηλά βρίσκεται η Κομισιόν λίγο βρίσκεται στα, στα, στα σύννεφα όσον αφορά το τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη και επίσης μας ανέφερε το ότι υπάρχει ένα κλίμα διακυβερνητικού τελείριου μεταξύ των κρατών μελών τα οποία προσπαθούν να συνοηθούν, να διασυνδεθούν με διάφορες, σε διάφορες ομάδες όμως ξεχνώντας την ε, ενωτική προσπάθεια η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό όραμα. Αν λοιπόν ισχύουν αυτά και αν τη σήμερα ημέρα το κοινοβούλιο, να το πούμε αλλιώ, είναι η ατμομηχανή είναι η τελευταία λύση, η τελευταίος θύλακας αντίστασης στις προσπάθειες συρρήγνωσης της Ένωσης. Επομένως, αν όλα αυτά ισχύουν, τότε έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη ε, και καλούμεθα να τοποθετηθούμε για το ποια είναι η γνώμη μας για την προτινόμενη μεταρρύθμιση. Επίσης, ε, η ευθύνη αυτή είναι προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία μεριά έχουμε την ε, ευθύνη μας όσον αφορά την οικονομική συγκυρία, τις πιέσεις, την κρίση, τις αγορές. Από την άλλη μεριά όμως επίσης έχουμε και τον προβληματισμό για τόσο αφορά τις μελλοντικές συνέπειες που είναι δυνατόν να έρθουν οι συνέπειες αυτές κατόπιν μιας τέτοιας μεταρρύθμισης και το πώς θα πολιτευτεί η Ένωση. Το είπε ο κ. Μπρόκ ότι ο μηχανισμός προβλέπεται και α μην είναι τόσο ρητό από τη συνθήκη. Ούτε είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι ε, αυτό θα έχει συνέπειε ανησυχητικές για το μέλλον. επομένω, ε, το πιο βέβαιο είναι όμως ότι θα έχουμε τέτοιου είδους δυσάρεστε συνέπειε αρνητικές και όπως το κύριο Χάφνερ, Επίση θα πρέπει να δούμε πώ θα δοθεί μία απάντησε από αυτή την Επιτροπή τη δική μας που θα δώσει μία ουσιαστική απάντηση αποτυπώνοντας εκεί τις ανησυχίες του, τη γνώμη του για το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην ιδέα για το ότι η μεταρρύθμιση της συνθήκης είναι ένα βήμα προς την, οικονόμηση, την ε, οικοδόμηση μιας ε, αυθεντικής οικονομικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει αυτό το διάβημα να γίνει. Όμως, αποφεύγοντας, όπως είπε και ο κύριος Γκουαλτιέρη, αυτό το διάβημα να αποτελέσει πίσω γύρισμα. Γιατί αυτή είναι η λογία του Κοινοβουλίου. Στο να τοποθετηθεί και κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είπε ο κύριος Μπροκ, να ανταποκριθούμε έτσι και στην αναγκαιότητα και ταυτόχρονα να αποφύγουμε, όπως είπε ο κύριος Γουαλτιέρη, να κάνουμε αυτό το διάβημα να πισωγίζουμε. Και για αυτή τη δύσκολη προσπαθία μας έχουμε δύο προτάσεις στο, σε σχέση με αυτούς που έλαβα το λόγο προηγουμένω. Να πούμε κάτι για το Eurogroup, να πούμε κάτι για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Να πούμε κάτι για την οικονομική διακυβέρνηση. Να πούμε κάτι για το εξάμεινο, το επόμενο, στο οποίο θα ρυθμιστούν τα δημοσιονομικά και με ε, αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνδυάσουμε αυτές όλες τις μεταβλητές και με αυτά τα οποία θα διατυπώσουμε στην εκθεσή μας να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε τη θεσμική έγκλη στην Ένωση και έτσι να αποφύγουμε τη συρρήγνωση των αρμοδιοτήτων μας των θεσμικών στο μέλλον. Από την άλλη μεριά εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση η οποία διατυπώθηκε και δηλαδή σε κάποια συνάντησή μας, ίσως στις 17 του μηνός, στο Στρασβούργο ίσως, δεν αναφέρεται ποια ημερομηνία, να καλέσουμε τον κύριο Τρισέ, τον ε, Επίτροπο, τον Αρμόδιο για τα οικονομικά και επίσης να πούμε στους συνεισηγητές της νομοδότησης ή στους ε, συντονιστές ε, να πούμε να έρθουν ούτως ώστε να τα συζητήσουμε. Κάτι το οποίο θα βοηθούσε για το δικό μας έργο αλλά και τους εισηγητές ούτω ώστε να δουλέψουν πιο ολοκληρωμένα. Επίσης, όπως είπε ο κ. Μέντες θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με αυτή την έκθεση, το νωρίτερο δυνατόν και κατά προτίμηση για τις άντρε επόμενης να έχουμε μια πρώτη έκθεση και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούμε συγκεκριμένα να τα συζητήσουμε. Εγώ δεν είμαι φανατικός όσον αφορά με την τήρηση του χρονοδιάγραμματος. Όμως θα πρέπει να τηρήσουμε αυτά τα οποία θέσαμε. Και εάν χρειαστεί μέχρι τελευταία στιγμή να υπάρχει κάποια παράταση, να μπορούμε να δώσουμε παράταση στο διάγραμμα από την άλλη μεριά όμως, αν μπορούμε να το τηρήσουμε, αυτό το οποίο προτάθηκε, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλή ένδειξη του ότι δουλεύουμε όπω πρέπει στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Σόντεγκαρτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολλά επιχειρήματα ακούστηκαν και ήδη η συζήτηση είναι μακρά. Και βάσει των επιχειρημάτων και της συζήτησης καταδεικνύονται δύο πράγματα. Είναι προφανές ότι αυτό που θα αποφασίσουμε είναι σημαντικό. Δεν είναι κάτι αδιάφορο ή κάτι απλό. Δεύτερον, είναι προφανές ότι ό,τι αποφασίσουμε θα διαγράψει μία πορεία για το μέλλον. Είναι κάτι το οποίο θα έχει μεγάλη επίπτωση, μεγάλη σημασία στα επόμενα χρόνια. Και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όσον αφορά την ίδια τη λειτουργία της Ένωσης. Στα πλαίσια της ομάδας μου, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω συζήτηση έτσι ώστε να εμβαθύνουμε στο ζήτημα. Από ό,τι κατάλαβα, οι άλλες ομάδες έχουν δεχτεί την απλουστευμένη διαδικασία και απέρριψαν την ε, πρόταση μιας ε, εντελεχέστερης συζήτησης και αυτό με λυπεί. Για πρώτη φορά η απλουστευμένη διαδικασία δεν μας προσφέρει καμία εγγύηση, όπως λέει και ο εισηγητής, ότι θα είναι πιο γρήγορη. Θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές τροποποιήσεις στη διάρκεια της συζήτησης ε, όπως έγινε και όσον αφορούσε το, τη συζήτηση ε, για τη συνταγματική συνέλευση. Είτε το θέλουμε είτε όχι, δημιουργούμε ένα προηγούμενο αυτή τη στιγμή εάν πιστέψουμε ότι αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας θα λύσει τα προβλήματα σταθερότητας του ευρώ, τότε απατώμεθα. Δεν ισχύει αυτό. Θα υπάρξουν νέες ανάγκες για αυτό το μηχανισμό σταθερότητας και τότε θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Την τελευταία φορά θα μας πούνε, θα μας πούνε λοιπόν τότε, μα την προηγούμενη φορά δεχτήκατε την απλωστευμένη διαδικασία, γιατί δεν δέχεστε τώρα. και επομένως η διαδικασία που ονομάζεται διαδικασία γενικής ε, μεταρρύθμισης ε, θα μετατραπεί σε διαδικασία απλουστευμένης μεταρρύθμισης. Αναθεώρηση, συγγνώμη. και τότε θα αναθεωρούμε διαρκώς όλα τα θετικά στοιχεία της συνθήκης της Λισαβόνας. Τι κάνουμε λοιπόν. Νομίζω τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη τη ομάδα μου, θα πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε να έχουμε μία σε βάθο συζήτηση. Και δεν πρέπει να είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι επειδή διαλέγουμε την απλουστευμένη διαδικασία αυτή θα είναι και μια γρήγορη διαδικασία. Θα δημιουργήσουμε απλώς ένα προηγούμενο. Θέλω να ζητήσω λοιπόν στους συζητητέ να γράψουν σαφέστατα ότι είναι η τελευταία φορά που δεχόμαστε την γρήγορη απλουστευμένη διαδικασία και ότι την επόμενη φορά οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω διασκέψεως γιατί διαφορετικά θα μας πιέζουν και θα μας εκβιάζουν διαρκώς. Και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του πότε θα πάρουμε απόφαση στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στο Στρασβούργο ή θα πρέπει να περιμένουμε 15 μέρες μετά για να πάρουμε την απόφαση στο, στις Βρυξέλλες. Και καλά τα λέει ο Άντριου Ντάφ. Είμαστε εδώ, έχουμε εκατοντάδες κάμερες ε, και, και, και τελικά έχουμε αποφάσεις του Κοινοβουλίου ε, τις οποίες ε, στέλνουμε στο Συμβούλιο, συνοδεία της αστυνομίας ε, κτλ. Μα εντάξει, αυτό είναι και λίγο θέατρο. Εάν το Κοινοβούλιο δεχτεί την απλουστευμένη διαδικασία έτσι κι αλλιώς, εάν όλες οι ομάδες με εξαίρεση τη δική μας έχουν δεχτεί το άρθρο 136 για τις διαδικασίες που προτείνεται τότε γιατί να κάνουμε τόσο θέατρο ας είμαστε ειλικρινείς Πρόεδρος, τρέχει τρέχει ο χρόνος, έχουμε μονάχα μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Βλέπω ακόμα τους Μορέιρα, Σόλπ, ε, Τέινεν και βεβαίω θα πρέπει να αφήσουμε και αρκετό χρόνο για του δύο ομιλητές, θα, τους δύο εισηγητές, συγγνώμη. Θα κλείσω λοιπόν με αυτούς τους τέσσερις ομιλητές και να τους παρακαλέσω να μην ξεπεράσουν τα τέσσερα, άντε πέντε λεπτά ε, ο καθένας. Ωραία Ιραήλ πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλές από τις ενστάσεις που ακούστηκαν και από αυτά, με αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκοτχέρη, αλλά η θεσμική αναθεώρηση των συνθήκων θα πρέπει, κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε τι είναι ρεαλιστικά δυνατόν, να βρούμε μια ρεαλιστική λύση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα που ανακύπτουν. Είναι απαραίτητο να λάβουμε αποφάσεις. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό, αλλά το κατά πόσον θα πρέπει αυτό να κατοχυρωθεί μέσω ε, τροποποίηση τη συνθήκη, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, δεν υπάρχει ρήτρα ε, ευελιξία ή ε, ενισχυμένη συνεργασία, δεν υπάρχουν άλλε δυνατότητε. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ένα τέτοιο μηχανισμό, ιδιαίτερα επειδή αμφιβάλλουμε και για την νομική βάση για τις άλλες ε, λύσεις. Αν υπάρχει λοιπόν ε, γίνει ε, ρητά και ανοιχτά αυτή η αλλαγή, ίσως να υπάρχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση τώρα για τον, τον χαρακτήρα τον διακυβερνητικό. Κοιτάξτε, είμαι φεντραλιστής. Το να αποδεχτώ έναν ε, κυβερνητικό μηχανισμό, ξέρετε, με δυσκολεύει λίγο. Αλλά ξέρουμε ότι αν ήταν αρμοδιότητα κοινωτική θα είχαμε αύξηση των κοινωτικών ε, αρμοδιοτήτων. Αυτό είναι σαφές. Οι διακυβερνητικοί μηχανισμοί, οι ευρωπαϊκοί κοινωτικοι μηχανισμοί. Θέλω, θέλω τέτοιους μηχανισμούς, γιατί πολλοι από τα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρειάζονται οι πιο αδύναμες χώρες. Δεν μου φαίνεται ότι υπάρχει συνέπεια, συνοχή με την νομισματική ένωση, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει να αποδεχτώ ότι είναι μια επιλογή το να υπάρξει ένας διακυβερνητικός μηχανισμός. Ο άλλος, η άλλη επιλογή είναι να μην κάνουμε τίποτα. Ε, από τα δύο αυτά επιλέγω λοιπόν το διακυβερνητικό ε, μηχανισμό για την απλοποιημένη διαδικασία. Υφίσταται, υφίσταται ήδη στη συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί. Οι αλλαγές αυτές, οι τροποποίησεις δεν χρειάζεται να γίνονται έτσι πάντα. Γιατί ξέρετε, εδώ στο σημείο αυτό σημαντικός είναι και ο χρόνος, ο παράγοντας του χρόνου. Όσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να αντιμετωπίσουμε τη δυσπιστία των αγορών. Το οποίο καθαστά ακόμα πιο ευάλωτε στις ευάλωτες χώρες. Και μετά υπάρχει και η διαδικασία επικύρωσης αν θέλουμε να επικυρωθούν αυτές οι αλλαγές, να ακολουθήσουμε την απλουστευμένη μέθοδο. Και έτσι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πολιτικό μέσο για να επιταχυνθεί η διαδικασία επικύρωσης και σε εθνικό επίπεδο. Άρα, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά και πολιτικά επιχειρήματα, για τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του μηχανισμού αυτού, κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό γίνεται μόνο μέσω της συνθήκης. Αν λοιπόν είναι η μοναδική λύση που έχουμε στη διάθεσή, σας, στη διάθεσή μας, ας το κάνουμε και το συντομότερο δυνατόν μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κ. Σόλτς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί με έχουν καλύψει πολλοί συνάδελφοι. Να πω το εξή. Το είπε και ο συνάδελφος Μπρόκ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Και αντίθετα με πολλούς συναδέλφους, πιστεύω ότι η κρίση δεν έχει ακόμα πάρει τέλος. Και στις ε, ευρωεκλογέ θα κληθούμε όλοι να εξηγήσουμε τι κάναμε, τι κάναμε προκειμένου να διαμορφώσουμε δομές πιο βιώσιμες, μηχανισμούς πιο αποτελεσματικούς τα τελευταία πέντε χρόνια, τα οποία θα αποτρέψουν τη συνέχιση και την όξυση της κρίσης. Άρα ανακύπτει το εξή θέμα και είναι δικό μας καθήκον να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών μας. Θα μας ρωτήσουμε λοιπόν πώς θα αναπτύξουμε μηχανισμούς τις οποίες θα καταλαβαίνουν οι πολίτες, τους οποίους θα αποδέχονται και που θα επηρεάσουν με τέτοιο τρόπο την καθημερινότητά τους που θα κερδίσουν εμπιστοσύνη, θα, θα, θα εμπιστευτούν την ε, ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Άρα η πολιτική συζήτηση που γίνεται εδώ συνδέεται με τα συνταγματικά και θεσμικά ζητήματα πολύ στενά. Η πολιτική συζήτηση λοιπόν θα πρέπει να συνδεθεί με τη θεσμική αυτή συζήτηση. Γι' αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα. Αν συνοψίσουμε το τι ακριβώς επιθυμούμε, ήμασταν στην αντιπροσωπεία με τη, στη Μεγάλη Βρετανία και το ερώτημα είναι τι περιμένουν οι Βρετανοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν την ε, καθημερινότητά τους. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να εξετάσουμε και με αυτό το πλαίσιο, με, αυτό αυτή τη σκέψη να ελέγξουμε τους μηχανισμούς μας. Ξέρουμε ποιε είναι οι πλειοψηφίε, ξέρουμε ποια είναι η στάση του Συμβουλίου γιατί θέλει να περάσουν τα συμφέροντά του. Ξέρουμε ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε μια πολιτική απάντηση των μελλοντικών θεσμικών αλλαγών. Δεν θα πρέπει να αποφύγουμε αυτά που συζητήσαμε και χτες. Την μεγαλύτερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη ακολουθώντας την συμβουλή σας και την επιθυμία σας. Ε, πολλά έχουν υποθεί από τους προλαλήσαντες συναδέλφους, ε, των οποίων συμμερίζομαι τα σχόλια και την επιχειρηματολογία. Νομίζω ότι εδώ στη Συνταγματική Επιτροπή αλλά και γενικότερα στο Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ε, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Αίσθημα ευθύνης το οποίο θα ακολουθείται όμως ε, και από την αίσθηση της πραγματικότητας και από τον ορθολογισμό, τον πραγματισμό και την αίσθηση ότι αντιμετωπίζουμε κάτι πολύ σημαντικό σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η απλουστευμένη διαδικασία νομίζω ότι εξηγείται λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιπέσει πολλές χώρες ε, της ε, ζώνης του ευρώ η κοινή γνώμη των ε, χωρών μας δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Τουναντίον θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να αναλάβουμε γρήγορη και αποτελεσματική δράση. Τώρα, το να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα με ε, ορθολογισμό ε, και αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μας αποτρέψει από το να σκεφτούμε και κάποιες άλλες ευρύτερες επιπτώσεις πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση ε, θέτοντας και το δικό μας λιθαράκι στο μελλοντικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πώς συμβάλλουμε λοιπόν ε, σε αυτό το οικοδόμημα, γιατί πολύ συχνά τα μηνύματα είναι ε, λίγο ασαφή. Ε, ποια είναι λοιπόν η πραγματική, η συγκεκριμένη έννοια που δίνουμε στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, ε, ποια είναι, ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο, ποιοι είναι οι άξονες μιας στενότερης οικονομικής συνεργασίας που μπορούμε να δημιουργήσουμε, ποια είναι τα εργαλεία, τα νέα καινοτόμα ας πούμε εργαλεία τα οποία θα μπορούσαμε να σφυριλατήσουμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ε, μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και άρα αποτελεσματικότερη πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε το πρώτο βήμα το οποίο θα πρέπει να μας ε, οδηγήσει σε πιο συνολικές ε, ε, επιλογές και που θα τις βρούμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι ο συντονισμός με τα εθνικά κοινοβούλια διαφαίνεται απολύτως ζωτική σημασία. Μιλάμε για οικονομική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, ίσως, ίσως στο μέλλον δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική αυτά πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να στηρίξω ανεπιφύλακτα ε, την πρόταση του Πρόεδρου Λαμασούρ για μια ε, συνολική διάσκεψη για τον προπολογισμό και θα πρέπει το Κοινοβούλιο μας να συμμετάσχει ενεργότατα σε αυτήν τη διάσκεψη. Ευχαριστώ. Τελευταία παρεμβαίνουσε η κυρία Τάινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Μπροκ, εν συντομία, για το κατά πόσο συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι συγητές να περιγράψουν εκτενώς την κατάσταση και να κάνουν και μια προοπτική παρουσίαση του, της μελλοντικής κατάστασης για το πού θέλουμε να πετύχουμε. Θα ήθελα στην έκθεση να πραγματευτούμε ε, εκτεταμένα τις διάφορες εναλλακτικές ε, λύσεις που έχουμε, τις διάφορες νομικές βάσεις, να κοιτάξουμε και την, ε, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα μόνο να ζητήσω στην μελλοντική παρουσίαση της μελλοντική κατάστασης, όπου υπάρχουν διαφωνίες και για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, αυτό που ονομάζουμε στη Γερμανία ε, φρένο ε, χρέους, απαγόρευση δηλαδή χρέωσης, να τα παρουσιάσουμε στην έκθεση με ανοιχτό αποτέλεσμα, χωρίς να προεξοφλήσουμε το αποτέλεσμα. Ιδάλλως η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να συγκεντρωθεί, την οποία επιθυμούμε βέβαια την πλειοψηφία αυτή. Θα δώσω τώρα στο λόγο, τον λόγο στους συγητάς έτσι ώστε να απαντήσουν και να αντιδράσουν στα επιχειρήματα που ακούστηκαν. Η πρότασή τους λοιπόν είναι το εξής. Να απαντήσουμε ναι ή όχι. Ή οποιαδήποτε και αν είναι η πρόταση, γιατί βλέπω ότι η κυρίαρχη τάση είναι για το ναι. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως να υπάρχει επιχειρηματολογία η οποία ε, να είναι πολύ συγκεκριμένη, να δηλώνει ότι εγγράφεται η διαδικασία αυτή σε μια πολύ γενικότερη διαδικασία. Ε, και έστω και αν όπως ακούστηκε, έστω και αν πρόκειται για μια διακυβερνητική, ε, ένα διακυβερνητικό όργανο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θα ενέχεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ε, τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ σημαντικό θέμα και από αυτού θα πρέπει να τοποθετηθούν οι συγητές. Τι θα κάνουμε, ε, θα πάρουμε την απόφαση στην επόμενη ολομέλεια ή θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Επίσης, ε, θα θεωρούσαν σωστό να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση όπου θα συμμετάσχει και κάποιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και ε, ο Επίτροπο Αρμόδιο για τα Οικονομικά Θέματα, ενδεχομένω και κάποιοι συνάδελφοι από την ΕΚΟΝ. Ο συνάδελφο Γκουαλτιέρη πρώτα θα απαντήσει. Λοιπόν, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκερέρο. πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο σημαντικές και σοβαρές ευθύνες. Πρώτον, η δύσκολη οικονομική κατάσταση και επομένως ε, την ε, ανάγκη με υπεύθυνο τρόπο να απαντήσουμε. Έχουμε απέναντί μας τις αγορές, έχουμε απέναντί μας χώρα σε δυσκολία, αλλά έχουμε και την ε, ε, υποχρέωση, έχουμε και αυτήν την ευθύνη ως ε, μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων να διασφαλίσουμε το συνταγματικό μέλλον της Ευρώπης. Επομένως, περιπλέκεται λίγο το θέμα Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι η ουσία είναι σημαντική και όχι το αβ ή γ ε, άρθρο. Και εγώ αναρωτιέμαι εάν δεν είναι πολύ σημαντικά τα θεσμικά θέματα ε, και μόνο ο ορθολογισμός και ο πραγματισμός ε, πρέπει να παίρνει το, το πρώτο χέρι, τότε τι έννοια έχει να έχουμε μια επιτροπή πολιτικών, συγγνώμη, συνταγματικών υποθέσεων. Και άλλωστε, ε, εμείς δεν είμαστε ένα δικαστήριο εδώ, εμείς είμαστε ένα πολιτικό όργανο το οποίο ασχολείται και με ε, ε, θέματα συνταγματικά. Ενδεχομένως μερικές φορές είναι ανιαρό να το επαναλαμβάνει κανείς, αλλά έτσι κι αλλιώς εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να αρκεστούμε στην ε, γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ όσον αφορά την τεχνική ουσία δεν πρέπει να δώσουμε απλά ένα ναι ή ένα όχι σε μια διακυβερνητική διάσκεψη. Βρισκόμαστε απέναντι σε μια απλουστευμένη διαδικασία η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς επ' αυτού θα δώσουμε μια γνωμοδότηση που δεν είναι δεσμευτική. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν να καθησυχάσω τους συναδέλφους ότι μπορούμε να δείξουμε όποιο βαθμό υπευθυνότητα, αλλά όσο μεγάλος και αν είναι αυτός ο βαθμός δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Σύμφωνα με τις συνθήκες η γνώμη μας δεν βαραίνει ιδιαίτερα. Επομένως θα κάνουν αυτό που θέλουν σχετικά με το μηχανισμό σταθερότητας. Εμείς απλώς πρέπει να εκφράσουμε μια γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενεργοποιήσει την απλουστευμένη διαδικασία βάσει της προτάσεως της βελγικής κυβερνήσεως και αφού θα έχουμε εμείς γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο και όχι μια επόμενη διακυβερνητική θα πάρει την απόφαση να τροποποιήσει τη συνθήκη της Λισαβόνας που θα τεθεί σε ισχύ ε, βάσει των συνταγματικών ε, συμφωνιών των 27 χωρών. Αυτό είναι με μεγάλη σαφήνεια αυτό που πρέπει να κάνουμε που καλούμαστε να κάνουμε. Από αυτή την άποψη δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει η γνωμοδότησή μας να αφορά ένα ναι ή ένα όχι. Ούτε μας ζητούν αυτό, ούτε ε, και η δικιά μας προδιάθεση είναι αυτή. Δεν, ε, το, κοινοβούλιο δεν, ε, δεν εκφράζεται δεσμευτικά με ένα δεσμευτικό ναι ή ένα δεσμευτικό όχι. Το, ε, το κοινοβούλιο πρέπει απλώς να γνωμοδοτήσει, λαμβάνοντας υπόψη και το μέλλον της Ευρώπης όχι ε, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ε, και τις ευαισθησίες κάποιων κοινοβουλίων. Ε, ωραία, να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Πολύ ωραία. Αλλά να είμαστε και υπεύθυνοι. Και επομένως... Ε, εάν πρέπει να καταπιούμε κάτι πολύ άσχημο, να μην χρυσώνουμε το χάπι και να λέμε τι ωραίο που είναι, δεν είναι καραμέλα με γεύση φρούτου αυτό που μας ζητούν να καταπιούμε Τώρα, το κοινοβούλιο, αν θέλει να γίνει πιο, ε, να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως ε, και να πει εγώ όχι, όχι, δεν θέλω καθόλου να ρίξω λάδι στη φωτιά, να μην εκφράσει το κοινοβούλιο την άποψή του όπως οφείλει, ε, πραγματικά βρίσκω ότι είναι κρίμα και για τους πολίτες που μας έστειλαν εδώ ακριβώς για να ελέγχουμε κάποιες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως, ναι, μεν μια επικοδομητική λογική και συμβιβαστική κατά κάποιο τρόπο πρόταση που δεν θα κλείνει όμως και εντελώς τα μάτια στην ε, συνταγματική πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω όπως λένε μερικοί άλλοι ότι η απλουστευμένη διαδικασία δεν είναι σωστή από μόνη της, ότι, θε, ότι χρειάζεται η διάσκεψη κτλ. Δεν είναι άποψή μου. Η απλουστευμένη διαδικασία μπορεί να είναι μια λύση. Εγώ απλώς θεωρώ ότι μπορούσαν να βρεθούν άλλες που παρουσιάζουν λιγότερο κίνδυνο, άρα μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι η πρόταση είναι σαφής. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να αναφερθεί αυτό σαφώς στη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Δεύτερον πρόβλημα, η ουσία. Για να αποσαφηνίσουμε καλύτερα τι σημαίνει διακυβερνητικό, μη διακυβερνητικό, εμείς βάζουμε στην, στις συνθήκες την αναφορά ότι δεν θα μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε αυτό, στο μέλλον αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός που δίνει χρήματα σε κράτη. και έχουμε τα 60 δις τα οποία ε, έχουν πρόθεση έτσι να ησυχάσουν τις ε, αγορές. Απ' την άλλη πλευρά όμως λέμε ότι δεν θα μπορέσουμε πλέον ποτέ αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αφαιρούμε κάποιες δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, για να ησυχάσουμε τις αγορές λέμε ότι ό,τι κάνουμε τώρα και ό,τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το 2013 είναι αντισυνταγματικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι η εξαιρετικότερη στρατηγική για να καθησυχάσουμε τις αγορές, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, αυτήν την, ε, ε, σε αυτή την αμαξιοστοιχεία κατά κάποιο τρόπο έχουμε μπει και πρέπει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ίδια μαξοστοιχεία. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να προτείνει έναν μηχανισμό στο εσωτερικό αυτής της διαδικασίας που θα μπορεί κατά κάποιο τρόπο όχι να βρίσκεται σε κοινοτικό επίπεδο. Εγώ έχω μία πολύ πιο μετριοπαθή πρόταση. Έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να ενταχθεί ε, στο μηχανισμό της ε, Ένωσης, παραμένοντας όμως για κυβερνητικός μηχανισμός. Όμως οι υπουργοί που θα πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα θα πρέπει να συνεδριάζουν στο Συμβούλιο. Γιατί ο, ο συνάδελφος Μάρτιν είπε ότι έτσι κι αλλιώς θα συντονίζει η Επιτροπή κτλ. Ναι, εντάξει, αλλά όλα αυτά δεν αναφέρονται, δεν γράφονται πουθενά. Δεν γράφεται στη διατύπωση την νέα της ε, συνθήκης και ούτε στην πρόταση της Επιτροπής και δεν ξέρω εάν είναι γραμμένα και στα ανεπίσημα κείμενα τα οποία συζητώνται. Επομένως, εγώ λέω ότι το Κοινοβούλιο, και συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει ο Μπρόκ, ότι το Κοινοβούλιο πέρα από την συνταγματικού περιεχομένου πρόταση θα πρέπει να ζητήσει να υπάρχει κάποια διασύνδεση ανάμεσα στο μηχανισμό αυτό ε, και την θεσμική έκφραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα λοιπόν από την γενική ευθύνη που φαίνεται ότι κανένας δεν την αναλαμβάνει τελικά. Πέρα λοιπόν από το να μην ε, δώσει κανείς τη γνωμοδότηση ε, και να ακολουθηθεί μια παρακολουτική ε, πολιτική στην οποία εγώ αντιτίθεμαι. Εμάς μας ζήτησαν και we have to deliver όπως μπορούμε να το πούμε απλά. Και θα πρέπει να πάρουμε την απόφασή μας πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική δέσμευση αυτή που αναλαμβάνουμε και στην ουσία ε, ε, ε, είναι το μόνο επί το οποίο δεν μπορούμε να πούμε όχι. Και, εν πάση περιπτώσει, στο χρόνο που μας απομένει, πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην εγγύηση του μέγιστου βαθμού ολοκλήρωσης ανάμεσα σε αυτό το μηχανισμό και τη θεσμική έκφανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο κύριος Μπροκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι μετά την εισηγήση του συνάδελφου Γκοτιάρη σχετικά σύντομο. Το μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στο πλαίσιο αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Και το να χρησιμοποιήσουμε το όπλο αυτό μας, μας δημιουργεί προβλήματα γιατί έχει και εξωτερικές συνέπειες. Άρα θα πρέπει και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να λάβουν την ευθύνη τους. Και τα περιθώρια λιγμού, τα οποία διακρίνουμε στο Συμβούλιο, να τα εξετάσουμε από πλευρά του Συμβουλίου, να δούμε τι μπορεί να λειτουργήσει. Κατά δεύτερον, διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι υπέρ του όχι. Τρίτον, τις προτάσεις για το τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνθήκη μου φαίνονται οι προτάσεις σας όλες πιο καλές από αυτές τις προτάσεις του Συμβουλίου και ιδιαίτερα αυτά που μας προτείνει και ο κύριος Ντάφος, εκπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης για το τι είναι δυνατόν να γίνει διαδικαστικά γιατί επίσης διαπιστώνω ότι υπάρχει και μια πλειοψηφία κατά της απλοποιημένης διαδικασίας. Α, εσείς είστε υπέρ, μάλιστα. Όλοι υπέρ είναι. Έχουμε τις προτάσεις Γκοτχέρη, την, το θέμα του αυτοματισμού, σε θέματα ελέγχου, σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθεροποίησης και ανάπτυξης, Πρόκειται για τροποποίηση της συνθήκης οι οποίες μπορούν να συμμορφωθούν, να συνάδουν με την ε, απλοποιημένη διαδικασία. Δεν έχω πιστεί, αλλά να είμαι, έχω ανοιχτό πνεύμα. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση όμως. ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την ενέργεια δημοψηφίσματος αν δεν υπάρχει ανακατονομή των αρμοδιοτήτων. Και αυτό είναι γεγονός. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε βρετανικό δημοψήφισμα να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, μια και πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν πλήττεται από την κρίση τη Ευρωζώνης. και όλα αυτά θα επηρεάσουν και την τελική μας τοποθέτηση για το ποια πολιτική οδό θα ακολουθήσουμε και τι προτάσεις θα, κατα... θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Καταγράψατε κάποια κοινά στοιχεία. Το 48-6 φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτό γιατί είναι προστευμένη διαδικασία. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ε, οι περισσότεροι ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία. Και 7 Φεβρουαρίου ε, θα πρέπει να έχουμε την, ε, την πρόταση έτσι ώστε 17 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο ε, να, να εμβαθύνουμε συγγνώμη, τη συζήτηση και ενδεχομένως να κάνουμε την ψηφοφορία 7 Μαρτίου στο Στρασβούργο ή 15 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και μετά να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια 9 Μαρτίου ή 24 Μαρτίου. Αλλά πιστεύω ότι το να ξανασυζητήσουμε μεταξύ μας στις 7 Φεβρουαρίου, εάν συμφωνούν οι συγητές, είτε είναι σε θέση είτε δεν είναι σε θέση να υποβάλουν μια γραπτή μορφή της έκθεσης νομίζω ότι είναι απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη την σημασία του θέματος. Εάν δε οι εισηγητέ ήδη την 7η Φεβρουαρίου είναι σε θέση να υποβάλουν ένα γραπτό κείμενο, οπωσδήποτε αυτό θα διευκολύνει κατά πολύ τη συζήτηση. Μέντες Δεβίγκο, θέλετε να πείτε κάτι. Συμφωνώ με αυτό το οποίο προτείνεται. Εδώ έχουμε δεσμευτεί και προ του ηγητέ να ακολουθήσουν αυτό το διαγράμμα. Και αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στα πρακτικά των συντονιστών. Επομένω, τι να σου πω. Δεν καταλαβαίνω γιατί να επιφυλασσόμεθα. Ε, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν για την εκθεσία, αλλά νομίζω ότι σήμερα ξεκάθαρα τοποθετηθήκαμε όσον αφορά το τι ρότα θα ακολουθήσουμε. Διάφορα μπορεί να γίνουν, τι να πούμε, τι τροπολογίες να κάνουμε για να μην χάνουμε χρόνο. Στις 24 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο. Στο τσακ θα το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το πρόβλημα. Τα ξέρουν οι εισηγητέ τα θέματα. Ε, Επομένω, να έχουμε το κείμενο προβδομάδα και έτσι θα μπορούσαμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ο επόμενο. Μουελτιέρη, όπως σας είπα, προσωπικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να σεβαστούμε το χρονικό περιθώριο της 24ης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο εργασία την επόμενη φορά. Ένα pre-draft. Ένα έγγραφο σαν αυτό που είχε υποβάλει ο συνάδελφος Μπροκ για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και επομένω μετά να έχουμε τη δυνατότητα ταχύτατα να προχωρήσουμε στο προσχέδιο. Επομένω, λέει ο πρόεδρο να έχουμε ένα γραπτό κείμενο. Ο συνάδελφο Μπρόκ ζήτησε να πάρει το λόγο. Πρόεδρε, να προγραμματίσουμε να τηρήσουμε το γρήγορο χρονοδιάγραμμα για να είμαστε άμεσοι στην αντίδρασή μα αλλά να κρατήσουμε και άλλες εναλλακτικέ λύσεις. Εγώ θα ήθελα προσωπικά προτού ολοκληρωθούν οι συζήτησει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και στη διάσκεψη των Προέδρων και στις συζητήσει που θα λάβουν χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να έχουν γίνει όλα αυτά. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει και με πέραν από αυτό θα γνωμοδοτήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να είναι ελεκτρωμένη εικόνα για τις γνωμοδοτήσεις αυτές προτού ε, ολοκληρώσουμε την άποψή μας και θα είχα να ολοκληρωθεί στις 8 του μηνός. Ε. Σας παρακαλώ να μας το επιτρέψετε αυτό. Θα πρέπει να είναι γρήγορη η διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγο να καθυστερήσουμε υπερβολικά. Εντάξει. Νομίζω ότι επομένως εδώ ζητούμε περισσότερη ευελιξία. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα νομίζω ότι μπορούν να γίνουν και περαιτέρω έκτακτες συνεδριάσεις, ας πούμε, την δεκάτη του μηνός. Και μετά θα έχουμε την δεκάτη εβδόμη. Άρα, να διατηρήσουμε, να, να γράψουμε στη μερίσια διάταξη την ε, δεκάτη, την ε, εβδόμη μάλλον ε, και να γράψουμε το ενδεχόμενο μιας έκτακτης στις 10 Φεβρουαρίου. Α, ναι, είχε προβλεφθεί ήδη η 17η Φεβρουαρίου, λέει ο Πρόεδρος. 14, 14 e Στις 14 μου λέει ο γραμματέας εδώ ότι ψηφίζει η ΕΚΟΝ. Ναι, θα, τρεις, τρία, λεπτά. Το, η ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ θα πάρει τρία λεπτά και δεν νομίζω ότι η ΑΦΚΟ δεν μπορεί ας πούμε να συνεδριάσει στο Στρασβούργο τη Δευτέρα το απόγευμα. Δεν θα μας αποτρέψει μία απλή ψηφοφορία να το κάνουμε. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο. Ωραία και αν μπορείτε να υποβάλλετε και ένα γραπτό έγγραφο. Να έχουμε. Γκουελτιέρη. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε και ε, περαιτέρω συζήτηση έτσι ώστε ε, πριν από το πραγματικό προσχέδιο να κάνουμε ένα πρώτο προσχέδιο, αυτό το pre-draft που έλεγα προηγουμένως. Επομένως, 7 και 14 Φεβρουαρίου. 7 και 14 Φεβρουαρίου. Και οι δύο άμεσα Συμφωνείτε 7 και 14 Φεβρουαρίου. Πάρα πολύ ωραία. Να σας υπενθυμίσω ότι για τις 7 Φεβρουαρίου έχουμε και ένα άλλο γρήγορο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μαθηματικής συνάντησης ε, στο Cambridge. Θα είναι ένα σημείο προς πληροφόρηση. Αυτά και πέρα στη συνεδριάσεως.